Okay, colleagues. The rapporteur for our first item, Frank Engel, wants to, has to go vote in another committee, so... Καλημέρα θα πρέπει κάποιοι να πάνε να ψηφίσουν σε άλλη επιτροπή. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε επομένως, για, με το 17, λέει η Πρόεδρος. Αλλά πρώτα-πρώτα θα πρέπει να πούμε καλώς όρισαν ε, τώρα μετά τις διακοπές κάποιοι συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθαν και είπαμε ότι έχουμε το θέμα του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου 2021 και συζητήσαμε επανειλημμένα το ότι τώρα η Επιτροπή έχει παρουσιάσει την πρότασή της για το επόμενο ε, πολιτές πλαίσιο και η Επιτροπή μας ήδη έχει εγκρίνει μια γνωμοδότηση ε, του Πολ Ρούμπιχ και επίσης για την εφαρμογή του EDF, του DCI, την ανθρωπιστική βοήθεια και σε εκείνα τα έγγραφα είπαμε ότι το νέο πολιτές πλαίσιο θα πρέπει να έχει κάποια μέσα ξεχωριστά για ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια και να μην υπάρξει περικοπή χρηματοδότησης. Όλα αυτά πριν την πρόταση της Κομισιόν. Τώρα που την έχουμε την πρόταση, προβλέπει, διαπιστώνουμε, έναν και μόνο κανονισμό NDICI ονομάζεται Neighborhood Development International Cooperation Instrument ολογράφος και καλύπτει και το DCI καλύπτει και το Ταμείο Γειτονίας και το EDF και το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας παραμένει ξεχωριστό συμφωνήθηκε δε με την διάσκεψη των Προέδρων να εκπονήσουμε σε συνεργασία με την ΑΒΕΤ μια έκθεση για αυτόν τον κανονισμό NDICI και έτσι να συμμετάσχουμε σε μια τέτοια ε, διαδικασία συναπόφασης. Και θα τον ελάβουν οι συνάδελφοι Έγγελ και Γκέρενς. Η Επιτροπή των Προπολογισμών είναι κυρίως αρμόδια επιτροπή και πρόκειται να συντάξει μία ενδιάμεση έκθεση που θα κατέβει στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο. Αυτά όσον αφορά την πρόταση για το MFR και ο δικός μας συγητής επ' αυτού είναι ο κύριος Έγκελ, ο κύριος Ρούμπιχ είχε αναλάβει την προηγούμενη, αλλά πρώτος ο Φρανκ θα λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ Λίντα και, ευχα... και συμπαθάτε με γιατί πρέπει σε λίγα λεπτά να φύγω να τρέξω στην ε, Λίμπε. Έχω μια ψηφοφορία ε, και ακριβώς την ώρα που προβλέπετε θα την κάνει ο Κλοντ Έχουμε μόνο λοιπόν σε αυτή την γνωμοδότηση που αφορά το πολιτές πλαίσιο και αφορά βέβαια την Επιτροπή μας, είναι λογικό, για αυτό το μέτρο διεθνού συνεργασία και πολιτική γειτνίαση. Δικά μα θέματα. Ακριβώς όπως είπες, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον συμφωνούμε με την ε, πρόταση της Επιτροπής. Αναφέρεται το ότι όλα θα καλυφθούν από ένα νομοθέτημα για το μέλλον. Καταρχήν συμφωνώ και το σχέδιο κειμένου μου αυτό το πνεύμα έχει. Οπότε λέμε ότι θα λάβουμε υπόψη αυτή τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτή τη νέα προσέγγιση θεωρούμε ότι θα είναι ευκολότερο να πετύχουμε τους στόχους μας. Έχουμε το άρθρο 208 της συνθήκης που αφορά την καταπολέμηση της φτώχεια. Επίσης, λέμε για το 0,7% όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια, τι θα πρέπει να υπάρχει στην περίοδο προγραμματισμού, την επόμενη. Επανειλημμένα έχουμε πει για το ότι θα πρέπει το Ταμείο Ανάπτυξης να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό Σχέδιο κειμένου είναι ε, σύντομο συνήθως. Ό,τι μπορούσα τα ανέφερα. Να τα συζητήσουμε συνάδελφοι και να δούμε τι τροπολογίες θα υπάρξουν. Πολλές από αυτές θα αφορούν αυτό το ε, εξωτερικό μέσο χρηματοδότησης. Α, άλλη προσέγγιση λέει η πρόεδρος η Ε, άλλη προσέγγιση είχαμε πριν την πρόταση για το νέο MFF. Συνάδελφοι, θέλετε το λόγο. Ο Σάρλ. Ο Κάραλος. Είσαι συνεισηγητής. Μπορείς να πάρεις το λόγο. Ναι. Είμαστε στην αρχή αυτού του Κολκοθά. Το σημαντικό είναι να επιτύχουμε τους στόχους που καταγράφονται και τεκμηριώνονται στη δογματική μας βίβλο, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη. Χθε είχα την ευκαιρία να σας υπενθυμίσω ότι είμαστε εξαιρετικά δυνατοί στις υποσχέσεις, αλλά όταν ε, έρχεται η ώρα να τις κάνουμε πράξη, βρίσκουμε ένα σωρό δικαιολογίες για να εξηγήσουμε την ε, ανικανότητά μας. Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί λοιπόν, καλύτερες επιδόσεις, καλύτερα στόχοπροσιλωμένοι, να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία. Δεν θα πρέπει τα μέσα να απειλούν το σκοπό τελικά και να ε, είμαστε δέσμοι των μέσων και να μην επιτυχάνουμε τελικά λόγω αυτού κανένα σκοπό. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, η ζεύρα τι είναι, άσπρο ζώο με μαύρες λωρίδες ή μαύρο ζώο με λευκές λωρίδες. Έχουμε δικλείδες ασφαλείας για να λύσουμε τα θέματα. Θέλουμε να έχουμε αποφασιστικότητα. Ή θα έχουν άλλες διαστάσεις οι πράξεις μας στην εξωτερική πολιτική και θα έχουμε εκεί άλλες δικλείδες ασφαλείας. Το θέμα είναι τι έχει περισσότερες πιθανότητες να δουλέψει. Τι απ' όλα, πιο απ' όλα. Το να εντάσσουμε όλα αυτά τα πράγματα στον προϋπολογισμό είναι μια διεκδίκηση που υπάρχει από τις απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά δεν τα έχουμε τηρήσει. Κάποια κράτη-μέλη εποφθαλμιούν και με ζήλια κοιτάζουν τα δικαιώματα που κάποιοι έχουν αποκτήσει ε, το δεύτερο ήμιση του προηγούμενου αιώνα και δεν θέλουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Εάν τώρα στο νέο εργαλείο, στο νέο μέσο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη πραγματικά ήταν μέρος αυτού, τότε θα άλλαζαν αυτά τα δικαιώματα. Δηλαδή, εντό του Συμβουλίου υπάρχει ένας πυρήνας που θέλει να υπερασπιστεί τα προνόμια του. Τα κράτη-μέλη δεν θα μας κάνουν κανένα δώρο σε εμά το Κοινοβούλιο. Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι, πρέπει να τα έχουμε συζητήσει επισταμένως μεταξύ μας, έτσι ώστε ε, να θέσουμε τους στόχους υπεράνω των ε, μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων που μας κάνουν τη ζωή πολύ περίπλοκη. Κατά τα λοιπά, ο Φράγκα είπε διάφορα πράγματα τα οποία με βρίσκουν απολύτω σύμφωνο και θα έχω και την ευκαιρία να επανέλθω ε, όταν θα συζητήσουμε τα επιμέρους θέματα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Θέλουν άλλοι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Νόιζερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως μπορούμε να συμφωνήσουμε στις ε, βασικές αρχές και προσεγγίσεις της γνωμοδότησης. Θέλουμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου, χωρίς όμως να εισέλθουμε σε σύγκρουση με τα εθνικά κοινοβούλια. Ο, δυστυχώς έχει φύγει ο Φρανκ Έγγελ, αλλά θα ήθελα να μάθω. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με αυτό που έχουμε ήδη συζητήσει και αποφασίσει στην Επιτροπή. Ποιες είναι οι διαφορές λοιπόν μήπως υπάρχει κάποια νέα γραμμή την οποία ακολουθεί ο Φρανκ Εγγέλ. Ο Παουλ Ρούμπικ έχει το λόγο ως συντάκτης προηγούμενης νομοδότησης. Νομίζω πως οι διαπραγματεύσεις για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα είναι ακόμα δυσκολότερες σε σχέση με το παρελθόν Υπάρχουν διάφορες νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και έτσι όπως ε, φαίνεται θα υπάρχει μια μεγάλη μειοψηφία ε, που θα διαφωνήσει με την ε, διάθεση του 0,7% του ΑΕΠ για αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε με, λεπτό, με περισσότερη προσοχή το πώς ε, θα δημιουργήσουμε ίδιους πόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς αυτό θα συνδεθεί με τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Στο μέλλον θα είναι πολύ σημαντικό αυτό για την αναπτυξιακή πολιτική, διότι πρέπει να έχει την ευκαιρία για προώθηση. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα απασχολήσει τους ε, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και δεν πρέπει να ξεχνάμε τι παίζεται. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο. Ε, να μιλήσω κι εγώ. Ο Φράγκα μίλησε για την ενσωμάτωση του ε, Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Βρίσκεται υπό έλεγχο το θέμα αυτό και σίγουρα το κοινοβουλευτικό έλεγχο του Κοινοβουλίου θα πρέπει να θεσμοθετηθεί στο νέο μέσο. Έχουμε κακό προηγούμενο ε, από το καλοκαίρι που μας πέρασε για τα δικαιώματα κοινοβουλευτικού ελέγχου του Κοινοβουλίου σε σχέση με τη συμφωνία με το Ιράν. Τα κρατη ειδοποιήθηκαν στις 11 ε, Ιουλίου. Εμείς δεν μάθαμε τίποτα, παρότι συνεδριάσαμε την ίδια ημερομηνία. Ε, μάθαμε μόλις στις 19 ε, του μηνός τι συνέβαινε και το συζητήσαμε χθε στην Επιτροπή. Επομένως, εφόσον ενσωματωθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, ναι, αυτό στην ουσία... Όντω προποθέτει δικαίωμα κοινοβουλευτικού ελέγχου από εμά, όμω δεν είναι και σίγουρο. Πρέπει να παλέψουμε για να το καταφέρουμε. Και νομίζω πως η θέση του Φρανκ Έγγελ είναι αρκετά διαφορετική από, την ε, προηγούμε, από τις προηγούμενες συζητήσεις και από αυτά που είχαν συζητηθεί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Σίγουρα πρέπει εντός των πολιτικών ομάδων να ε, υπάρξει μία σαφή στάση και ένα όραμα. Γι' αυτό πρέπει να συζητήσουμε με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Δεν έχει ζητήσει κανείς το λόγο, οπότε θα δώσω το λόγο. Α, όχι, Σάρλ, έχετε το λόγο. Να προσέχουμε να μην προβαίνουμε σε βιαστικά συμπεράσματα. Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας. Χθες ε, συνεδρίασαν οι τέσσερις συνεισηγητές και δεν απέδωσε και πολλά η συνάντησή τους. Να εστιάσουμε το ενδιαφέρον και την προσοχή μας στην πεπτουσία αυτού του εγχειρήματο, να πούμε ποιο είναι καλό για την ανάπτυξη, ποιοι είναι οι σκοποί μας και ποια είναι τα καλύτερα μέσα να πετύχουμε αυτούς τους σκοπούς. Και συμπληρωματικά, επικουρικά, από από ένα, για έναν παρατηρητή από ένα πολύ μακρινό πλανήτη υπάρχουν και ε, οι επιδιώξεις και τα προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, να να προβλέψουμε τέσσερι περιπτωσιολογικέ μελέτες. Δεν είναι δυνατόν το Κοινοβούλιο να μην έχει ένα δικαίωμα επίβλεψη στα κονδύλια που δίδονται για την ανάπτυξη. Η Εκομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αυτή που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Και αν δεν κάνουμε εμεί τη συγγραφή υποχρεώσεων για να τη πούμε πώ θα το διαχειριστεί, θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Τα δικαιώματα αυτά πρέπει να ενισχυθούν με μία προϋπόθεση. Η μελλοντική αρχιτεκτονική δομή της λήψης των αποφάσεων πρέπει να είναι έτσι ώστε η Κομισιόν να λαμβάνει υπόψη της τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή να πούμε ξεκάθαρα ότι ή θα έχουμε μία πλημμύρα εφαρμοστικών πράξεων, δεν ξέρω ε, ποιο άρθρο της συνθήκης σε έρχεται εκεί, 289 νομίζω, το 289, ή θα έχουμε κατεξουσιοδότηση πράξης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει δηλαδή να να υπάρχει ένα εργαλείο που να μας επιτρέπει να ασκήσουμε το βάρος μας και να το κάνουμε αισθητό το βάρος μας στους υπόλοιπους. Να ξεφύγουμε από την πεπατημένη και να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τη λειτουργία των αναπτυξιακών πολιτικών που εφαρμόζουμε, διατηρώντας και ενισχύοντας κιόλα αν μπορούμε το δικαίωμα επίβλεψης εξέτασης κοινοβουλευτικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα είναι εύκολο αυτό. Και σε μεταγενέστερα στάδια, από εδώ και μπρος, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την αντιπαράθεση, αυτή την αντιπαραβολή, ε, να αντιπαραβάλλουμε, να βάλουμε δίπλα-δίπλα αυτά που έχουμε προβλέψει και αυτά που εφαρμόζονται τελικά και αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Και πρέπει να έχει κανείς πολύ καλή θέληση για να τα εξετάσει με ψυχραιμία και να βγάλει το ζουμί και να δει τι μπορεί να βελτιώσει. Αλλά δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα πριν κάνουμε την ανάλυση. Είμαστε στην αρχή αυτή τη διαδικασία, δεν έχουμε ολοκληρώσει την ανάλυση μα. Πρέπει να έχουμε πολύ υπομονή και αποφασιστικότητα. Και θα πρέπει να βιαστούμε για να μπορούμε να έχουμε επιχείρημα στέρεο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Ε, είναι μια περίοδος που στρεσάρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ξέρω. Είναι ίσως η περίοδος που πιέζεται περισσότερο από όλες τι άλλε περιόδου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν θα αφήσουμε τα όπλα κατά μέρο. δεν θα παραδώσουμε τα όπλα. Έχουμε επιχειρήματα και θα πρέπει να τα προβάλλουμε. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Φέλιξ Φερνάντεθ Σόρ, Διευθυντή τη DG Τεύκο και Φίλιπ Μπέρντο Σεριάνη, δεν ξέρω ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος, ο Φέληξ σας. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Ε, οι περισσότεροι εξημών με ύψιλον που είπατε ότι είναι όντως μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρχεται στα καθημερινά της καθήκοντα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ε, Ευχαριστούμε τον εισηγητή, τον Φράγκ, για την επικοδομητική στάση που έχει υιοθετήσει κατά τη σύνταξη της γνωμοδότησής του. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια προσπαθώντας να αυξήσει το μέρος του προϋπολογισμού, της πρότασης προϋπολογισμού που ε, θα προορίζεται για την εξωτερική δράση. Αυξάνονται και τα κονδύλια ε, για την εξωτερική δράση και για την ανάπτυξη. Το έχουμε προβλέψει αυτό στην πρότασή μας στο 92% από το 90% που έχουμε σήμερα, 90% ως προς τα ODA και αυτό έχει σχέση και με αυτό που είπε ο κύριος Ρούιμπιχ, ότι όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της συνολική συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και για τον αντίκτυπο που θα έχει εξωτερική χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το έγγραφο που συντάξαμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Φεβρουάριο, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημόσια δηλώνει ότι προκειμένου να διατηρήσουμε το επίπεδο ε, φιλοδοξίας ε, εν ώψη του 2030 και το επίπεδο του 0,7 τότε η ποσότητα στόχος θα πρέπει να είναι τα 142 και όχι τα 123 και θα πρέπει να γίνουν κάποιες εξισορροπήσεις και αντισταθμίσεις εντός του σώματος των επιτρόπων και γι' αυτό καταλήξαμε στο νούμερο που βλέπετε που αποτελεί σημαντική αύξηση ούτως ή άλλως. Αυτό καταρχάς κατά δεύτερο λόγο. Τα τελευταία χρόνια, αν όχι και δεκαετίες, έχουμε μιλήσει για την ένταξη στο προϋπολογισμό, τον τακτικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ανάπτυξη. Ήταν πρόταση αυτό το 2011. Και εγώ ήμουν σε αυτή τη θέση, αλλά όχι σε αυτήν εδώ, στη θέση του Φιλιμπέρτο καθόμουν τότε. Αλλά φέτος το παρουσιάζουμε, το προτείνουμε, το υποβάλλουμε, το επιθυμούμε. Αυτό αυξάνει την κοινοβουλευτική παρουσία, την παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα, στα, της εξωτερικής δράσης και κατά 30%. Εάν το EDF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη, μπει στο τακτικό προϋπολογισμό όλες οι δαπάνες για τον Ειρηνικό, για την Καρυβική, για τη ΑΚΕ, για τις χώρες κάτω από τη Σαχάρα, την Υποσαχάρη Αφρική, το Σαχέλ, ε, θα είναι όλες αυτές οι δαπάνες στο τακτικό προϋπολογισμό με απότατο άρχοντα και αφέτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ε, αποφασίζει για αυτά τα κονδύλια. Τώρα, ακόμα και να πούν τα κονδύλια στο καταπιστευματικό ταμείο, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος της τακτικής διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Βλέπετε, αυτό δεν θα μπορούσε να έχει γίνει. Βλέπετε λοιπόν ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ακριβώς αυτή που επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να αυξήσει την εξουσία που έχει στη διαχείριση του προπολογισμού σε σχέση με το Συμβούλιο. Τέλος. Χαίρομαι που ακούω από εσά ότι ναι, οι προκλήσεις θα είναι μεγάλες, αλλά ε, το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ ασφικτικό. Είναι σημαντικός ο πολιτικός ρόλος του Κοινοβουλίου, ο ρόλος που θέλει το ίδιο το Κοινοβούλιο να ασκήσει και εξετάζοντας το χρονοδιάγραμμα και της δικής σας Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, βλέπουμε ότι οι εξελίξεις θα είναι θετικές και θα φτάσουμε τελικά στο σημείο που επιθυμούμε. Αλλά θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Φιλιμπέρτο, αν επιτρέπετε, γιατί έχει να προσθέσει κάποια πράγματα σημαντικά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Λίντα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και από τη δική μου πλευρά. Να πω κι εγώ με τη σειρά μου ότι βεβαίως και καλωσορίζουμε τον τόνο και την, ε, το ύφος του σχεδίου γνωμοδότησης το γεγονός ότι δίδεται έμφαση στο πώς αλληλοσυνδέονται οι διάφορες δράσεις, η εξωτερική δράση με την ανάπτυξη, με τη μετανάστευση, με την κλιματική αλλαγή. Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι ο εισηγητής έχει μια πολύ επικοδομητική στάση σε σχέση με το NDICI, το εργαλείο και το μέσο για την ανάπτυξη, τη γειτονία και την διεθνή συνεργασία. Έχουμε λοιπόν πόρους από, για την ανάπτυξη και το σχετικό ποσοστό που προτείνουμε. Η πλήρης προσθετικότητα, αθρηστικότητα των πόρων για να αντιμετωπιστούν πτυχές που δεν είναι αμυγός αναπτυξιακές. Αυτό είναι το βασικό. Συμφωνούμε με τον εισηγητή Θέλουμε να προστατεύσουμε και να αυξήσουμε τους πόρους για να στηρίξουμε τους στόχους της χιλιετίας και την ανάπτυξη γενικότερα και ε, να αντιμετωπίσουμε πολιτικές που, ε, προκλήσεις μάλλον, όχι πολιτικές, να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις που είναι διασυνδεδεμένες και είναι εγκάρσιες, άπτονται διαφόρων τομέων. Θέλουμε να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό και έτσι θα είμαστε σε θέση να αντιδρούμε γρήγορα σε νέες συνθήκες ή στη γεωπολιτική που τόσο ραγδαία εξελίσσεται σε διάφορα μέρη του κόσμου λόγω οικονομικών φορέων, παραγόντων, δημογραφικού, μετανάστευσης και νέων τάσεων, γιατί ξέρετε ότι σε πολλές περιοχές του κόσμου οι πολιτικές τάσεις είναι αρκετά ισχυρές και ε, μπορεί να υπάρξουν ε, σημεία καμπής. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε διασύνδεση για να μπορούμε να παίξουμε όλα τα χαρτιά της τράπουλας που έχουμε στο χέρι μας, να μην μένουμε μόνο σε ένα χρώμα. Και σε σχέση με αυτά που είπε ο Φέλεξ για τη συμπερίληψη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ανάπτυξη στον τακτικό ε, προϋπολογισμό, θα ήθελα και εγώ να πω αυτά που είπε ο Κρίστιαν επανειλημμένος εδώ, ότι δηλαδή είναι ανάγκη να προβληματιστούμε, να σκεφτούμε ποια εμπειρία έχουμε αποκομίσει από την παρελθούσα συνδιαλλαγή μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως για παράδειγμα το στρατηγικό διάλογο που έχουμε τα τελευταία χρόνια, για να είναι ο διάλογος συνεχής και να έχει νόημα. Να μην στρέφουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένα επιμέρους διοικητικά βήματα και χρονοτριβούμε εκεί. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοιχτή, επιθυμεί ιδιαίτερο να συζητήσει τρόπους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βελτιώσει ε, την ανταλλαγή απόψεων και τη συνεργασία ε, για να προσανατολίσουμε καλύτερα την εξωτερική μας δράση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Φρανκ Έγγελ δεν είναι εδώ για να απαντήσει, οπότε η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 30 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στις 9 Οκτωβρίου. Περνάμε τώρα στο σημείο 18, 24η διάσκεψη για την ε, Σύμβαση Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή COP24. Η διάσκεψη το 2015 ήταν ιδιαίτερα σημαντική και οδήγησε στην διαθέτηση ε, της Συμφωνίας του Παρισιού. Η εφαρμογή της ε, Συμφωνίας του Παρισιού τώρα πρέπει να περάσει σε ε, στάδιο ολοκλήρωση. Γι' αυτό λοιπόν προετοιμάζουμε μια πρόταση ψηφίσματος για να συνεισφέρουμε και εμείς στην, στο έργο της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει κάποια επίσημη διαδικασία, οι συντονιστές μας αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν την άτυπη διαδικασία του e-tray. Και να ακολουθήσουμε την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, προετοιμάζοντας ορισμένες τροπολογίες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον φάκελο που έχετε και στάλθηκαν στις πολιτικές ομάδες. Αυτές κατόπιν πρέπει να ορίσουν οι συγητές και μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου πρέπει να σταλούν οι τροπολογίες πίσω στην Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω δύο λόγια για τις τροπολογίες μου και να ζητήσω από τους συντονιστές να ενημερώσουν τους συναδέλφους ε, για το ότι πρέπει να μείνουμε εντός των ορίων της αρμοδιότητας της Επιτροπής μας και να μην τα ξεπεράσουμε. Διότι στο παρελθόν έχει συμβεί να μας ενημερώσουν άλλες επιτροπές ότι οι τροπολογίες μας αφορούν παιδεία της δικής τους αρμοδιότητας. Ορισμένα από αυτά τα θέματα εξετάζονται από τις τροπολογίες εδώ ε, και ίσως ε, κάποιος εκπρόσωπος της ε, Γενικής Διεύθυνσης Clear θα μπορούσε να μας ενημερώσει για ε, το που βρισκόμαστε σε σχέση με την χρηματοδότηση για την ανάπτυξη. Πριν έρθω στην Επιτροπή αυτή, ήμουν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και θυμάμαι ότι σε κάθε, μετά από κάθε κόπ κάναμε υποσχέσεις, είχαμε μεγαλοπίβολα σχέδια, αλλά οι υποσχέσεις αυτές δεν τηρούνταν στην ολότητά τους. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να έχουμε κάποια ενημέρωση σχετικά με το που βρισκόμαστε. Μετά, οι υπόλοιπε τροπολογίες έχουν ε, να κάνουν με τα βιοκαύσιμα. Υπήρξαν περιπτώσεις ε, στο παρελθόν σε ορισμένε από τις φτωχότερε χώρες του πλανήτη να ε, χρησιμοποιείται γη για την καλλιέργεια βιοκαυσίμων και να αναγκάζονται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να τις εγκαταλείψουν. Επίσης, οι τροπολογίες αναφέρονται στο ότι πρέπει να δοθεί ένα τέλος ε, στην χορήγηση πιστώσεων για τα ορυκτά καύσιμα. Και επίσης, ο Ντέιβιντ Μακάλιστερ, πρόεδρο Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και εγώ συναντηθήκαμε με την συντονίστρια των ΗΠΑ για την περιοχή του Σαχέλ και μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει έκκληση για επενδύσεις, επενδύσεις μικρής κλίμακας, ιδιαίτερα ε, σε αγρότες. πάνω από το 90% της ηλεκτρικής ενέργειας ε, διοχετεύεται στις πόλεις σε αυτές τις χώρες, αλλά το υπόλοιπο 10% που ζει στην Ήπεθρο αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες ηλεκτροδότησης ε, και δεν μπορεί να εργαστεί λόγω της έλλειψης ε, ηλεκτρικής ενέργειας. Το ζητούμενο λοιπόν, αυτή η έκκληση, είναι να γίνουν περισσότερες επενδύσεις στην παροχή ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και, τις, ε, και στην ύπεθρο αυτών. Αυτές είναι λίγο πολύ τροπολογίες που κατέθεσα. Έπρεπε να εργαστούμε γρήγορα διότι δεν είχαμε πάρα πολύ καιρό με τους χειώδεις εισηγητές, όμως ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συζητηθεί το θέμα περαιτέρω. Ε, ο Μπόγκταν έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, να πω ότι συμφωνώ με τη θέση σας και πράγματι βρισκόμασταν υπό χρονική πίεση. Έπρεπε να εργαστούμε πάρα πολύ γρήγορα. Όμως η θέση της Επιτροπής μας για την COP24 πρέπει να ε, παρουσιαστεί. Πρέπει να παρουσιάσουμε και τροπολογίες από τις πολιτικές μας ομάδες και παρότι γνωρίζω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο για να μπούμε σε λεπτομέρειες, νομίζω πως οι γενικέ γραμμές θα πρότεινα και εγώ να ακολουθήσουμε τις προτάσεις σου. Ευχαριστώ πολύ. Και μια που έχουμε σήμερα εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Γενική Διεύθυνση Κλίμα και από τη Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ, θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει φέτος, για το πώς ε, πάνε τα πράγματα. Και θα δώσω τώρα τον λόγο στην ε, κυρία Λίνα Μπάρτζα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Η COP24 πράγματι πλησιάζει. Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από το Παρίσι και από τότε οι διαβουλεύσεις μας είχαν επίκεντρο βασικούς στόχους. Καταρχάς, όπως αναγνώρισε και η πρόεδρος ε, Μακάβαν, στόχος είναι να συμφωνήσουμε για τους ε, κανόνες του Παρισιού, για τις ε, μεθόδους και τους τρόπους ε, διακυβέρνησης έτσι ώστε τα συμβαλώμενα μέρη να αποκτήσουν εμπιστοσύνη ε, στη... στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη-μέλη. Ε, εδώ πρόκειται για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα διέπει την συμφωνία για το κλίμα. Ο δεύτερος βασικός στόχος είναι ο διάλογος, ο οποίος ε, θα ε, διευκολύνει στην ε, συγκέντρωση πληροφοριών σε έναν απολογισμό, αν θέλετε, για το τι έχει γίνει στα τρία χρόνια που πέρασαν από το Παρίσι, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν από τους ηγέτες στην COP21. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε αρκετά καλή θέση, μπορεί να ηγηθεί και στους ε, δύο τομείς. Η πρόταση για την διακυβέρνηση είναι πάρα πολύ καλή και θα είναι απόλυτα συμβατή με τους νέους κανόνες. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να μοιραστούμε την εμπειρία που έχουμε στον χώρο αυτόν ο στόχος του 40% τουλάχιστον ε, είναι σε καλό δρόμο. Έχουμε σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο. Πριν το καλοκαίρι ήδη έχουμε ε, καταφέρει να ε, συμφωνήσουμε σε πολλά που μας βάζουν σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων για το 2030. Επίσης, οι εταίροι μας, ιδιαίτερα οι οικονομίες του G20, οι εκπομπές των οποίων αναλογούν στο 8% των παγκόσμιων εκπομπών έχουν συμφωνήσει για ε, τους ε, για εξίσου φιλόδοξους ε, στόχους και έχουν δεσμευτεί για την ανάληψη δράσης. Και σε πολιτικό στάδιο ο διάλογος ε, θα παρέχει την ε, ευκαιρία να γίνει αυτό. Η επόμενη φάση του διαλόγου θα λάβει χώρα στο Κατοβίτσε της Πολωνίας. Θα συνεισφέρουμε, λοιπόν, στο ψήφισμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος μέσω των τροπολογιών, ε, διότι με αυτόν τον τρόπο θα συνεισφέρουμε σημαντικά στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κλιματική αλλαγή, σε τελική ανάλυση, είναι μια τεράστια πρόκληση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Δεν μπορείς να μιλήσεις για την ανάπτυξη χωρίς να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και το αντίστροφο. Οι στόχοι λοιπόν και των ε, δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν είναι πανταχού παρούσα και έχει πλήξει ιδιαίτερα τις ε, πιο ευάλωτες χώρες και αυτές που είναι λιγότερο έτοιμες, ε, Αφρική, Καραϊβική, χώρες του Ειρηνικού. Όπως ήδη αναφέρθηκε λοιπόν, η χρηματοδότηση για το κλίμα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του, της Συμφωνίας του Παρισιού. Είναι μια ένδειξη αλληλεγγύης έτσι ώστε να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν αυτό που αναπόφευκτα έρχεται και να επιτύχουν επίσης ε, τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την ενεργειακή αυτάρκεια που φυσικά συμφωνούν και με τους ε, στόχους για το κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει αναλάβει δράση, έχει επιτύχει πολλά. Υπάρχει η πρωτοβουλία για την ενέργεια, η πρωτοβουλία για την ηλεκτροδότηση στις χώρες Αφρικής που έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο. Επίσης, ε, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προκλήσεις στην εφαρμογή των νέων ε, έργων και μεθόδων, όμως νομίζω πως ε, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και με τις άλλες χώρες δωρητές ε, για την έβρεση λύσης. Οι ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας δεν είναι μόνο πρόκληση για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και για ε, τις ανεπτυγμένες οικονομίες, τη βαριά βιομηχανία που εξαρτάται από αυτή. Είναι λοιπόν κάτι που απασχολεί όλους. Επίσης υπάρχουν οι δεσμεύσει της ε, Κοπενχάγης, τα 100 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020 που θα κινητοποιηθούν και από δημόσιους και από, ε, και από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Η δέσμευση αυτή έχει αλλάξει η πορεία από τότε που ένας από τους ε, μεγαλύτερους δωρητές άλλαξε τη στάση του. Συνεχίζονται βέβαια οι διαβουλεύσεις θεωρούμε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες, το G77 δηλαδή, κατανοούν απόλυτα τις επιπλοκές που προκύπτουν από την απόφαση μιας πολύ ισχυρή κυβέρνηση να αλλάξει τη στάση της. Θα πολλαπλασιάσουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας και θα προσπαθήσουμε έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, αλλά και από την πλευρά των ε, ε, χωρών που λαμβάνουν τη βοήθεια. Μετά, χρειάζεται να αυξηθεί η προβλεψιμότητα και η διαφάνεια. Αυτό είναι, είναι δύο από τους ε, σημαντικούς στόχους του Κατοβίτσε. Ε, αυτά από μένα προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση, λέει ο Πρόεδρος. Δεν συζητάμε τα θέματα του κλίματος ε, αρκετά. Νίκολα για τραντώνει από την Ρωτούμε Δούμε, θα πρέπει τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νέα προγράμματα, τα νέα μέσα και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει κατάλληλη προκοδότηση για τα έργα τα οποία πρόκειται να βοηθήσουν το θεματολόγιο για την επόμενη περίοδο, δηλαδή μέχρι το 2030 και έτσι να δούμε τι θα γίνει και με τους ε, βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. σε σχέση με τη συμμετοχή των Παρισίων για να δούμε τι λέει η Ντεύκο. Εσείς τι κάνετε για την ΚΟΠ. Ας πούμε, γιατί μπορούμε να τα πούμε με όλους τους πρέσβεις, τους εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σωστά είπατε, κυρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Και θυμάμαι πριν από πάρα πολλά χρόνια πήγα στην ε, Κένια και είδα εκεί πω έχει κατάσταση. Τι γίνεται με τις βροχέ του γεωργού που θέλανε βοήθεια, σπόρους. Οι οποίοι φυσικά οι άνθρωποι ήταν προετοιμασμένοι για τα δυσκολότερα, αλλά θα πρέπει να καλύψουμε και εκείνον τις δραστηριότητες στα προγράμματά μας. Άρα θα πρέπει κάτι να κάνετε ε, στη, στην πράξη και να δούμε πώς όλα αυτά θα μπουν στον προγραμματισμό. Antonio, please, the floor is yours. Good morning. First of all, I'm very sorry for my impossible surname. I know it's very difficult. Συμπαθάτε με. Ναι, το επώνυμό μου είναι δύσκολο, δύσκολο για όλους. Πιέτρα Αντώνη ονομάζομαι, πυρετό στην ΤΕΒΚΟ, στην Μονάδα για την Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια κλπ. Να απαντήσω σε αυτά τα οποία είπατε και να συμπληρώσω την Ελίνα. Πρώτα-πρώτα, χρηματοδότηση, μετάφραση των δεσμεύσεων, του προγραμματισμού, Όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να έχουν πρακτικό αντίκρισμα, αλλά θα πρέπει και να χρηματοδοτηθούν. Και στην ΤΕΒΚΟ κάνουμε τώρα μια αξιολόγηση για το τι γίνεται με τη χρηματοδότηση, να δώσουμε 20% του προπολογισμού για το κλίμα. Ε, έτσι και προχωράμε. Έχουμε το στόχο του 20% λοιπόν, 14 με 17 τα στοιχεία μας λένε ότι 19% ήταν ο στόχος και το πετύχαμε και δώσαμε 6,37 δις. Αυτά ε, τώρα δαπανώνται. Βέβαια υπάρχει διαφορά μεταξύ δέσμευσης και ε, δαπάνης γιατί αλλάζουν κάποια πράγματα διαχρονικά οπότε βλέπουμε ότι η τάση είναι ανωδική όσον αφορά την πρικοδότηση που διατίθεται και ταυτόχρονα Νομίζω ότι τα προγράμματά μας ε, είναι πετυχημένα. Ε, υπάρχει επομένως ε, τομιακή υποστήριξη του προϋπολογισμού και σε πολλές χώρες αναπτυσσόμενες έχει καταστεί πολύ σημαντικό ζήτημα συνεργασίας το κλιματικό. Ανεβαίνει, ανεβαίνει σε, στις προτεραιότητες. Και από πλευράς Ένωσης Έχουμε τα 100 δις που έχουν δεσμευθεί. Σε αυτά αναφέρθηκα πριν. Άρα έχουμε πρόοδο προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το πώς οι υποσχέσεις θα γίνουν πράξη, πολύ βασικό είναι το να έχουμε συντονισμό με τα χρηματοοικονομικά μέσα. NDC και η Συμφωνία των Παρισίων να ληφθούν υπόψη. Πολύ σημαντικά είναι τα εξή τρία στοιχεία. Το μισό των πόρων που έχουν δαπανηθεί για το κλίμα είναι θέματα προσαρμογής. Ιδίω οι φτωχότερε χώρε να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Άρα κάποια μέτρα που να μετριάσουν στην πρώτη φάση τα θέματα και φτάνουμε μέχρι το 55% σε συνολικές δαπάνες. Άλλο σημαντικό. Αυτά τα μέτρα συγκράτησης, μετριασμού είναι θέματα που μας απασχολούν και στο μέλλον όλες οι χώρες ε, θέλουμε να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια των NDC. Θέλουμε να πετύχουμε τα εξής δύο επίσης το πώς θα εμπλέξουν τον ιδιωτικό τομέα. Σωστά αναφέρατε την χρηματοδότηση από την Τράπεζα Επενδύσεων. Μόγλευση για αυτές τις παροχές προς τις χώρες και ταυτόχρονα αυτό το blending που όλο ένα και πιο σημαντικό είναι στη συνεργασία με τις χώρες εκείνες. Και άρα είναι σημαντικό το ταμείο που θα κάνει τη μόχλευση να είναι του ιδιωτικού τομέα. Και οι υπολογισμοί να είναι ρεαλιστικοί. Πολλές φορές βλέπουμε υπέρ αισιόδοξη στάση από τους δωρητές. Θα έπρεπε να είναι πιο προσγειωμένοι. Και η μεθοδολογία αντιστοίχως θα πρέπει να είναι λογική. Όλα αυτά αντιστοιχούν στις υποσχέσεις μας βέβαια. Και όταν μιλούμε για την προσαρμογή, όπως γνωρίζετε, έχουμε μία σειρά πρωτοβουλειών παγκοσμία ε, ε, εμβέλειας. Έχουμε τις κυβερνήσεις, έχουμε άλλους εμπλεκόμενους, όπως οι τοπικές αρχές, κοινωνία των πολιτών, ιδιωτικός τομέας, Έχουμε τη Συμμαχία για την αλλαγή του κλίματος. Αυξήθηκε η α, ε, πρικοδότηση. Έχουμε τον, την πλατφόρμα των δημάρχων. Επομένως, έχουμε και από τη βάση ανάληψη δράση, όχι μόνο από την κυβέρνηση. Γι' αυτό και η χρηματοδότηση προβλέπει για όλους πάροχες Βεβαίως και θα τα συζητήσουμε εδώ για να δούμε πώς θα σχεδιαστούν τα μέσα ε, συνεργασίας και αν χρειαστεί θα ψάξουμε και άλλα στοιχεία. Πρόεδρος. Βεβαίως και θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν στα νέα μέσα και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτό το 20%. ουσιαστικό τρόπο δηλαδή να καλύψουν στις πολιτικές μας την αλλαγή του κλίματος και όχι μηχανιστικά. Δεν έχουμε επίσημη διαδικασία, άρα ούτε και επίσημη προθεσμία για τροπολογίες. Άρα ό,τι προτάσεις έχουν ε, οι πολιτικές ομάδες να τις στείλουν στην ε, γραμματεία μας. Θα τα εντάξουμε όλα αυτά στο κείμενο. Αν προκύψει προθεσμία θα σας πω γραμματεία. Θα πρέπει μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας να σταματήσουν, να ολοκληρωθούν οι επαφές των πολιτικών ομάδων και να δούμε εάν θα θεωρηθεί απαραίτητο να οριστεί κάποια προθεσμία. Πάντως 24 Σενάτου είναι η συνάντησή μας, ε, μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθεια. Να προβληματιστούν επομένως μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, λέει η Πρόεδρος τότε θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το οριστικό κείμενο για να υποβληθεί. 6 Σεπτεμβρίου, επομένω, Παρασκευή. Θα υπάρξει χρόνο να συζητήσουμε στο Στρασβούργο για το συμβαστικό συνετικό κείμενο. Πάμε στο 19 τώρα, συνάδελφοι. Είχαμε προσθέσει στη μέση διάταξη δύο θέματα γιατί συνεχίζεται η ανθρωπιστική κρίση από ό,τι μαθαίνουμε σε δύο χώρες. Και άρα πρέπει να ενημερωθούμε για τα θέματα που έχουν ανακύψει. Έχουμε και εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ. Okay, yes, we have, we have, we have the DG Echo here. So, so, colleagues, we've discussed Gaza before. Ήδη έχουμε ξανασυζητήσει για την Γάζα. Και με την UNRWA, την ανθρωπιστική κατάσταση που ξέρουμε ότι είναι ανησυχητική και στη λωρίδα της Γάζας γιατί υπάρχει θέμα ασφαλείας, κλείσιμο συνόρων. Κρίση που επιδεινώνεται. Εμείς είμαστε εταίρος σημαντικός των Παλαιστινίων, της Παλαιστινιακής Αρχής και επίσης συνεργαζόμαστε με την UNRWA και έχουμε επίσης τη ΣΥΠΑ που συνεργάζονται. Μπορείτε να μας ε, ενημερώσετε, κυρία Βαλεντίνα Ντεμπερνάντη, που ασχολείστε με την Μέση Ανατολή. Έχετε το λόγο. Καλημέρα και ευχαριστούμε που μας καλέσατε με την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη Γάζα. Είμαι τελείο Ιουνίου για να σας πούμε τι γίνεται. Τι εξελίξεις είχαμε στο τελευταίο δίμηνο. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε ε, τώρα χαρακτηρίζεται από ηρεμία αλλά εύθραυστη. Μπορεί να γίνει όμως ε, ε, η έκρηξη ανα πάσα στιγμή. Είχαμε ένταση και βία αρχάς Αυγούστου και μόνο σε μια νύχτα της 8ης 8 8 πάνω από 50 πυράβλους προς το Ισραήλ ε, και η απάντηση ήταν 40 στόχοι που επλήγησαν. Σκοτώθηκαν τέσσερις άμαχοι, ε, ένα παιδί, μία έγκυος. Οπότε ήταν κρίσιμες αυτές οι στιγμές και θεωρούσαμε ότι θα ξεσπάσει η ανοιχτή αντιπαράθεση. Τώρα έχουμε κάθε Παρασκευή εκεί στο, στο τείχο, στο φράχτη έχουμε διαδηλώσεις τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε μικρές ομάδες που συγκεντρωνόντουσαν εκεί ανταλλαγή πληροφορισμών εκεί οι τραυματισμοί αυξάνονται κάθε μέρα και από τα τέλη Μαρτίου που έγινε τότε η μεγάλη πορεία 177 ήταν οι νεκροί Παλαιστίνοι και 19.000 οι τραυματίες. Απλώς των εξελίξεων του θέρους είχαμε απαγορεύσεις για την διακίνηση, για την πρόσβαση στα βασικά περάσματα. Κλείσανε μεταξύ 19 και 27 8. Αυτό για να πάρετε μία ιδέα. Το, το Ράφα προς την Αίγυπτο είχε κλείσει μια εβδομάδα, τώρα ξανά άνοιξε. Περίπου 300 είναι οι Παλαιστίνοι που κάθε μέρα θέλουν να πάνε στην Αίγυπτο. Και από αυτούς τους 300-200 περνάνε με βοήθεια της, ε, του Αιγυπτιακού συντονισμού, έτσι το λέμε, δηλαδή ότι θα πρέπει άτυπα να καταβάλουν 150 δολάρια, μεγάλο είναι το ταξίδι προς την Αίγυπτο και βέβαια τους ψάχνει πάρα πολύ προσεκτικά η Αιγυπτιακή ε, αστυνομία, το ίδιο όσον αφορά τα εμπορεύματα και εκεί το καλοκαίρι τα πράγματα ήταν ε, προβληματικά ανοιξε 15 15-8 πλήρω. για πρώτη φορά ε, επί ένα μήνα. Είχε κλείσει 9 εβδόμου ε, από για κάποια καύσιμα κατεπήγοντα και φάρμακα. Όλα τα άλλα εμπορεύματα δεν περνούσαν. Τίποτα δεν επιτρεπόταν να μπει ε, ούτε με τον διαγωνισμό ανασυγκρότηση του 14. Επομένω όλα είχαν κλείσει. Στις 17 εβδόμου επίσης είχαμε καύσιμο και ε, αέριο και λοιπά. 24 Εβδόμου επίσης επιτράπει να υπάρξουν κάποια καύσιμα κατεπήγοντα και αυτό στις 15 Αυγούστου οπότε είχαμε τρία ναυτικά μίλια μόνο ε, που αυξήθηκαν στα 9 για το ψάρεμα. Αυτό σημαίνει ότι όλο το καλοκαίρι δεν μπορούσαν οι ψαράδες να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους και η σημερινή κρίση που κράτησε όλο το 18 αλλά τώρα έχουμε αυτή την κορύφωση και τελευταίο δίμηνο είναι το θέμα του, της ηλεκτρικής ενέργειας. Τον Αύγουστο ήταν σταθερή η παροχή αλλά μόλις 4 ώρες κάθε μέρα. Όλα αυτά για το Ισραήλ ο μόνος πάροχος κάτω από 20 ΜΒ την ημέρα. Οπότε η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη. Στις 28 ο συντονιστής είπε ότι θα πρέπει η κοινότητα να χρηματοδοτήσει καύσιμα. 4,5 εκατομμύρια δολάρια χρειάζονται ούτως ώστε να υπάρχουν οι βασικότερες υπηρεσίες να λειτουργήσουν μέχρι το τέλο του έτους. Σας δώσουμε μια ιδέα τώρα ο ΙΕ Μήπως μπορείτε να τα λέτε πιο αργά, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν οι διερμηνείς για τη μετάφραση. Υπάρχει, υπάρχει χρόνος. Όλα αυτά τα νούμερα μπερδεύουν την κατάσταση. Όπως αναφέρατε κι εσείς, είχαμε περίπου όλοι εξαρτώνται από τα καύσιμα που τώρα τα παρέχει ο ΙΕ. Οπότε τώρα δεν υπάρχουν καύσιμα και αυτό έχει επιπτώσεις όσον αφορά τις βασικές παροχές υπηρεσιών υγιεινής, υγείας, τα νοσοκομεία ε, για τους γεννήτριές τους, μόνο ότι δορίζεται. Όταν είναι μόνο τέσσερις ώρες η παροχή του λιγού μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται. Τώρα Τελειώνει η τελευταία δόση της δωρεάς καυσίμων του ΟΗΕ και από το τέλος του μηνός δεν θα υπάρχουν καύσιμα. Οπότε θα έχουμε περίπου 4.800 ασθενείς που τώρα εξαρτώνται από ηλεκτρικές συσκευές και τα νεογέννητα ε, θα θέλουν βοήθεια. Και επίσης έχουμε ε, χιλιάδες άλλων ασθενών που θα πληγούν αν δεν υπάρχουν καύσιμα. Όπου καταλαβαίνετε όλα αυτά είναι κατά επίγουσης ε, επίσης, να σας δώσουμε εδώ τώρα μια ιδέα πού είναι το πρόβλημα. Βλέπετε δύο σημεία διάβαση για τους ε, ε, ανθρώπους και για τα εμπορεύματα. Δεξιά βλέπετε τα γραφήματα για την κατάσταση Βλέπουμε πάντω στο πρώτο γράφημα ότι υπάρχει μια βελτίωση σχέση με το 17. Παρ' όλα αυτά όμως παραπλανά λίγο αυτό το γράφημα γιατί το 17 ήταν η χειρότερη χρονιά όσον αφορά την ελευθερία διακίνησης. 51% λιγότερη από το 16 τότε. Οπότε έχουμε βελτίωση αλλά πάλι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όσο θα έπρεπε. Οπότε έχουμε τους ε, εκπρόσωπους κοινότητα, κοινότητας, όλο όλοι πρέπει να μετακινηθούν, οπότε δεν αρκεί αυτό. Ε, και στο Κέρεμ Σαλόμ βλέπετε επομένω ότι η τάση είναι καθοδική. Τον Αύγουστο ήταν κλειστό το Σάλομ, άρα η τάση πάλι θα είναι αρνητική. Επίσης ένα άλλο στοιχείο, ίσως σας ενδιαφέρει, αφορά τις ιατρικές εξετάσεις Όσοι θα πρέπει να πάνε σε γιατρό εκτός της ζώνης πρέπει να περάσουν από την ζελνή ασφάλεια. Έχουμε 245 που θέλαν να το κάνουν αυτό και εγκρίθηκαν 25%, 38% ε, απορρίφθηκαν. Το 38% είναι αύξηση σε τον προηγούμενο μήνα αρχές του 18. Είναι πολύ υψηλό ποσοστό και είναι πρόβλημα. Οπότε όσον αφορά αυτή την παραπομπή των ασθενών για μια απόφαση δικαστηρίου του Ισραήλ κατόπιν τεσσάρων οργανώσεων ανθρωπιστικών και τώρα, έλεγε το δικαστήριο, θα πρέπει να αφήνουν οι Ισραηλινές αρχές να πάνε από τη Γάζα ασθενείς έξω, σε γιατρό. Υπήρχε πρόβλημα με τη Χαμάς όσον αφορά κάποιες οικογένειες που είχαν σχέση με την οργάνωση, οπότε μέχρι τώρα να, να ληφθεί αυτή η απόφαση από το δικαστήριο δεν επιτρεπόταν σε και σχέση με τη Χαμά να πάει σε γιατρό εκτός ζώνη. Τώρα βλέπουμε συνδυασμένο αποτέλεσμα όλων αυτών των ε, πάρα πολλών τραυματιών. Έχουμε επίση άλλους περιορισμούς όσον αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων προ τα μέσα και προς τα έξω και ισορρευμένο αποτέλεσμα είναι αυτό στο ότι έχουμε όλες αυτές τις ε, ανθρωπιστικού χαρακτήρα ε, ανάγκες. δεκάδες χιλιάδων και δεξιά μπορεί να δείτε την ανάλυση ανά ηλικία, και βλέπετε πόσοι έχουν χτυπηθεί από πυρά και σύμφωνα με τον ΟΗΕ μέχρι τα μέσα Ιουλίου 59% των τραυματιών ε, είχαν πυροβοληθεί στο κάτω μέρος του σώματος στα κάτω άκρα και όσον αφορά το MSF στη Γάζα αυτοί οι τραυματισμοί ήταν ε, εξαιρετικά σοβαροί και πάρα πολύ δύσκολο να θεραπευθούν και έτσι οδήγησαν σε αναπηρίες. Πρέπει να περάσουν από χειρουργείο επανειλημμένα αυτοί οι άνθρωποι, φυσιοθεραπεία και αποκατάσταση. Ε, ακροτηριασμοί, επίσης να λεφθούν υπόψη το ότι έχουμε ε, μολύνσεις 20% των ε, τραυματιών και ίσως ε, και άλλο 40% και αν γίνει αυτή η επιμόλυνση, επιμόλυνση, τέλος πάντων υπάρχει πρόβλημα κροτηριασμού Άρα το σύστημα υγείας καταραίει και δεν αφορά μόνο εμάς τώρα, αλλά και το, το μέλλον, για τους αυριανούς, γιατί ε, ούτε καν με τώρα άμεση βοήθεια θα το πρόβλημα. Άρα δυναμητίζονται και οι μελλοντικέ προσπάθειες για τη Γάζα. Άρα χρειάζεται εξειδημένο προσωπικό, το δε Ιούλιο 40% των βασικών ε, φαρμάκων είχαν εξαντληθεί, 48% σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας ε, είχαν μόνο ένα μήνα ε, υλικό και όλα αυτά μέσα Ιουλίου συνολικά. Από τα τέλη Μαρτίου περίπου 7.500 Είχαμε 7.000 χειρουργία που αναβλήθηκαν. Πάρα πολλοί ήταν οι ασθενείς, δεν υπήρχαν κλίνες, στα νοσοκομεία δεν υπήρχε ηλεκτρισμός. Και στα νοσοκομεία εκεί την Τετάρτη διώχνουν τους ασθενείς γιατί περιμένουν νέου ασθενεί ε, την Παρασκευή και όταν τους διώχνουν ενώ ότι διώχνουν έναν ασθενή ανεξαρτήτως του πώς σοβαρή είναι η κατάσταση. Έχουν γίνει παλιμένες επισκέψεις από παντού και επομένως είπαμε για την ηλεκτρική ενέργεια που επηρεάζει άμεσα το αν υπάρχει καθαρό νερό, αν υπάρχει συνθήκες υγιεινής. Δεν μπορεί να πιει κανείς το 97% του νερού στη Γάζα, αλλά θα πρέπει να αγοράσει κανείς το νερό ή να το ζητήσει από διεθνή οργανισμό. Επόμενη κατάσταση επικίνδυνη από πλευρά ε, υγείας αλλά και περιβάλλοντος για, από τα λίμματα που πάνε στη θάλασσα. Εκατομμύρια είναι αυτά τα λίμματα τα οποία κάθε μέρα ε, εκατομμύρια λίτρων λιμάτων κάθε μέρα. Κρίση ρευστότητας επίσης. Πέφτει η αγοραστική αξία και αυξάνεται ο αριθμό των φτωχών οικογενειών. Σύμφωνα με την Παλαιστινική Στατιστική, τέλος του έτους είχαμε 53% φτωχού στη Γάζα από το 38,8% του 11%. Άρα πάνω από τους μισούς στην Γάζα χαρακτηρίζονται ως πέννητες. Η ανεργία 42%. Αν κανείς όμως ε, δει τι γίνεται, με τους ε, νέους που έχουν ε, κάνει κάποιες σπουδές πάμε στο 60%. Επομένως, συνολικά όλα αυτά είναι πολύ ανησυχητικά. Να σας δώσω μια ιδέα της απόκρισης της διεθνούς κοινότητας από πλευρά ανθρωπιστικής που καλύπτουμε τα δύο τελευταία χρόνια 540 εκατομμύρια δολάρια βλέπετε ότι ακόμα χρειάζονται περισσότερα. Και επίσης έχουμε μια λευκή βίβλο πλευρά που ζητεί 43,8 εκατομμύρια δολάρια Μάρτιο με Δεκέμβριο για να σωθούν ζωές κυρίως θέματα υγείας σε σχέση με όλους τους τραυματίες που έρχονται. Ακόμα λείπουν 21 εκατομμύρια μέχρι τον Δεκέμβριο η Ιούνορβα, όπως ξέρετε, βοηθάει. Τελείωσαν τα λεφτά τον Ιούνιο για τα κατεπήγοντα, οπότε τώρα θα πρέπει να βρεθεί χρηματοδότηση. Αυτά για να καταλάβετε τι γίνεται. Πνευματική υγεία, προγράμματα για απασχόληση. Λείπουν ακόμα 45 εκατομμύρια για την Παλαιστίνη και κυρίως για την Γάζα. Άλλα δύο εκατομμύρια για ανάγκες εκτός Ούνρουα. Παρακαλώ. Για να δούμε την ε, ανταπόκρισή μας από πλευράς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε 20 εκατομμύρια το 17 Το 19, 24 εκατομμύρια. Για τη Γάζα τα περισσότερα και λέμε για το πώς τώρα θα υπάρξουν και άλλα. Προτεραιότητες παραμένουν οι ίδιες, τα είπαμε. Υγεία, υγιεινή, έτοιμη για καταστάσεις ανάγκες αλλά έχουμε κάνει πισωγύρισμα από την οικοδόμηση ανεκτικότητος στην αντιμετώπιση των κατεπλούτων. Όλα αυτά επομένως ε, για να 46 εκατομμύρια φέτος. Και σας ευχαριστώ. Thank you very much. You paint Σας ευχαριστώ πολύ. Μας ε, σκιαγραφίσατε μια πολύ οδυνηρή ε, απεσιόδοξη εικόνα για την ανθρωπιστική κατάσταση, η οποία ήδη ήταν δύσκολη. Από τότε όμως που αναζωπηρώθηκαν οι διαμαρτυρίες για το ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε αναγνώρισαν την μεταφορά της πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ, και έπραξαν με αυτόν τον τρόπο, η κατάσταση όντω έχει επιδεινωθεί. Ξέρουμε από την Ούνρα τι περικοπέ στον προπολογισμό του, αλλά δεν είναι το πρόβλημα μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι και να φτάσει η βοήθεια και να μπορέσει να μπει μέσα στη λωρίδα τη Γάζα. Η κατάσταση είναι πραγματικά ε, πολύ κακή. Και ευτυχώ έχουμε τη Μάρκρετ Άλκρεμ, που είναι αντιπρόεδρο τη αντιπροσωπεία τη κοινοβουλευτική για τι σχέσει με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Όχι, ε, κάνω λάθος, τα διαβάζω και τα διαβάζω λάθος. Δεν μπορέσατε να πάτε στη λωρίδα της Γάζας, Μάρκαρετ, έτσι δεν είναι. Έκανα λάθος, τα διάβασα λάθος. Εσείς θα πάρετε το λόγο και θα μας πείτε... Μιλούμε για τα ανθρωπιστικά ζητήματα σε αυτήν την Επιτροπή. Γι' αυτά θέλουμε να μας πείτε. Ναι, αλλά συνεχίζουμε να είμαστε και πολιτικό κόμμα. Δεν είμαστε ανθρωπιστικός φορέας. Πρέπει να μιλήσουμε και πολιτικά. Επομένως, ναι. Δεν μπορέσαμε το DPAL να πάει στη Λόριδα της Γάζας από το 2009 ή το 10 είχαμε πάει μέσω χάφα και από τότε μας αρνούνται την πρόσβαση. Δεν είναι αποδεκτό αυτό. Το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να μιλήσει με πιο ισχυρή φωνή να ασκήσει πολύ πιο έντονη κριτική για το γεγονό ότι δεν μπορούμε να πάμε. Ξέρω κάποια πράγματα γι' αυτά και μπορώ να πω ότι στηρίζω αυτά που λέει η ΕΚΟ. Η κατάσταση είναι καταστροφική και θέλω να προσθέσω και το εξής. Βασική ευθύνη είναι το Ισραήλ με τα κατεχόμενα και την πολιορκία, τον αποκλεισμό της περιοχής αυτής, γιατί αυτό ε, ε, υπάρχει. Και υπάρχουν και κάποιες ευθύνε για την Παλαιστινιακή Αρχή. Πρέπει να το πούμε και αυτό βέβαια. Αλλά, εν περιπτώσει, δεν είναι αποδεκτό να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση με, το, με τον ηλεκτρισμό, με το φυσικό αέριο, ε, ως άσκηση πολιτικής πίεσης, ως πολιτικό μέσο. Και το Σεπτέμβριο όταν πάμε θα το θέσουμε ε, στο θέμα στην ΠΑ, στην Παλαιστινιαρική Αρχή, γιατί δεν θέλουμε να βλέπουμε τέτοια πράγματα. Ναι, πρέπει να αυξηθεί η βοήθεια γιατί η κατάσταση είναι δραματική. Να θυμόμαστε όμως το βασικό κανόνα βάσει του οποίου δίνουμε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει η ανθρωπιστική βοήθεια να μετατραπεί σε αναπτυξιακή βοήθεια, γιατί αλλιώ δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης. Δεν, η δυνατότητα ανάπτυξη δεν υπάρχει όχι λόγω κάποια φυσική αιτία π.χ. σεισμού, αλλά λόγω τη πολιορκία, του, του αποκλεισμού, του εμπάργου. Όλα είναι κλειστά, δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, οι επιχειρήσει δεν μπορούν να προμηθευθούν. Ε, όλα έχουν σταματήσει, έχουν παραλύσει. Άρα κρατάμε τη λωρίδα της Γάζας σε χειρότερη κατάσταση δίνοντας τους ανθρωπιστική βοήθεια. Τους κρατάμε σαν ζώα μέσα σε κλουβί και συζητάμε πόσο, ε, πόση τροφή χρειάζεται να τους πετάμε μέσα στο κλουβί και πόσο συχνά χρειάζεται να το καθαρίζουμε. Αυτό είναι τελείως απαράδεκτο. Ε, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να μπορούν να έχουν πρόσβαση, να πάνε στη Λωρίδα της Γάζας και να δουν την κατάσταση. Και χρειαζόμαστε και πολιτική βούληση, για παράδειγμα από την κυρία Μογκερίνη. Η Μογκερίνη έχει προσαρμόσει αυτή την ιδέα ότι υπάρχει και ευθύνη της Αιγύπτου και της Χάφα. Δεν πρέπει να ε, αφήσουμε τα πράγματα σε αυτό το μοντέλο τάχα, σύμφωνα με το οποίο τάχα το Ισραήλ έχει αφήσει τη λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο. Δεν είναι έτσι, δεν ισχύει αυτό. Είναι μέρος των Παλαιστινιακών εδαφών, πρέπει να ε, συνδέονται αυτά τα δύο μέρη και μπορούμε να ασκήσουμε πολύ μεγάλη πίεση. Δεν μιλάω για τιμωρίες ούτε για κυρώσεις θα επιβάλαμε κυρώσεις οποιοδήποτε άλλον εκτό του Ισραήλ αν συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο, αλλά θα αφήσουμε αυτό κατά μέρο. Τέλος πάντων, έχουμε πολιτικά μέσα στη διάθεσή μας και η, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποια μέσα. Άρα, ναι, να δούμε τη Συμφωνία εταιρική Σχέσης, άρθρο 2 πρέπει να το αναφέρουμε παραβίαση ανθρωπιστικών νόμων, καταστρατήγηση αυτών. Αυτό συμβαίνει Άρθρο 2 στη Συμφωνία Εταιρική Σχέσης είναι ένα νομικό μέσο, αλλά και εδώ έχουμε απευθύνει έκκληση για αληθινή διαφοροποίηση, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει να κάνει μόνο με το Ισραήλ και όχι με τα κατεχόμενα ε, εδάφη. Δεν είναι μόνο το θέμα ε, της ε, σήμασης κάποιων προϊόντων της ετοκετοθεσίας τους, αλλά θα πρέπει να, να έχουμε όλες τις επικοινωνίες απρόσκοπτες και αυτό, είναι, αυτό γίνεται για να εφαρμόσουμε τους δικούς μας νόμους και τις δικές μας αποφάσεις. Είναι ντροπή να δεχόμαστε να μην το κάνουμε στην περίπτωση της Παλαιστίνης και είναι εξωφρενικό όταν βλέπει κανείς τι γίνεται στη λωρίδα της Γάζας. Και Δεν ξέρω πότε ήταν το τελευταίο ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να ε, απευθύνουμε έκκληση για τη στρατηγική διαφοροποίηση. Και το εγκρίναμε αυτό με πλειοψηφία. Και στα Ηνωμένα Έθνη το Δεκέμβριο του 2016 έχουμε το 2334 που αναφέρεται σε αυτό το μέσο ως μοντέλο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε ούτε καν τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για, ως εργαλεία ως μοχλούς για να πετύχουμε το σκοπό μας. Άρα ποια εξοπιστία έχουμε. Χρησιμοποιούμε τα μέσα μας για άλλες περιπτώσεις και άλλες χώρες και βρίσκουμε μέχρι και κυρώσεις μάλιστα και εδώ είμαστε απλά ε, ε, σαν κυριούλες και λέμε σας παρακαλούμε στο Ισραήλ μήπως να τους δώσετε λίγο περισσότερη τροφή, μήπως να τους δώσετε λίγο περισσότερα φάρμακα, μήπως να ανοίξετε λίγο την πόρτα να πάρουν ελάχιστο αέρα, δεν είναι αποδεκτό αυτό. Πρέπει η κυρία Μογκερή να εθετήσει μια πολύ πιο ισχυρή στάση. Είναι δραματική η κατάσταση. Πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας και στη Παλαιστίνη που προσπαθούν να κινητοποιήσουν ε, τα πλήθη για μια μη βίαιη αντίσταση. Είναι αφόρητο το ότι δεν εγείρουμε αντιρρήσεις ε, σε αυτή τη μάχη που κάνει το Ισραήλ ενάντια σε άοπλους ανθρώπους που διαμαρτύρονται γιατί βρίσκονται υποκατοχή και υποπολιορκία. Ουσιαστικά στοχεύουν πολίτες. Και λέμε συνέχεια για το Ισραήλ ότι είναι ο καλύτερος μας φίλος και η πιο δημοκρατική χώρα της περιοχής και το καθεξής. Θα πρέπει όμως να κάνουμε πολύ περισσότερα. Έχουμε τα μέσα, την ισχύ αλλά και την ηθική υποχρέωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε ε, για αυτά που μας είπατε. Ο Ενρίκε Γκερέρο Σαλόμ είναι μέλος της αντιπροσωπείας και πηγαίνει στην Παλαιστίνη και είναι εκπρόσωπος της Επιτροπής μας για την ανθρωπιστική βοήθεια. Όταν επιστρέψει λοιπόν θα έχει διεξάγει διάλογο με την Παλαιστινιακή Αρχή για τα ζητήματα που αναφέρατε. Σίγουρα θα συναντηθεί με την Ούνρα και με άλλες οργανώσεις. Να προσθέσω όμως το εξής, λέει η Πρέπει να επενούμε την Ούντρα, γιατί ο λόγος για τον οποίο πράγματι αξίζει να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα υπάρχει Παλαιστινιακό κράτος είναι και η Ούνρα ε, έτσι ώστε όταν υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος αναγνωρισμένο να μην ε, αλληλοφαγωθούν μεταξύ τους και να καταστραφούν όλα. Η Ούνρα κάνει μια τρομερή εκπαίδευση στους νέους ανθρώπους στη Γάζα και βεβαίως πρέπει να ε, φτιάξουμε σχολεία. Το τσιμέντο μπορεί να χρειαστεί για να φτιάχνονται οι σύραγγε υπόγειε επικοινωνία, αλλά χρειάζεται επίσης και για να χτίζονται σχολεία. Η Ούνρα κάνει μια εξαιρετική δουλειά, αλλά έχει εξαντληθεί με αυτόν τον τρόπο ε, αντιμετώπισης από τις Ενωμένε Πολιτείε, αλλά και από ορισμένου εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ε, συνεχούν, συνεχίζουν να αποκαλούν αυτούς τους κατοίκους ε, πολίτες τρομοκράτες. Ο κύριος Έλλη θέλει το λόγο. Συμφωνώ απόλυτα δεν έχει νόημα να δίνουμε κι άλλα χρήματα για αναπτυξιακή βοήθεια όταν συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, όταν οξύνεται μάλιστα αυτή η κατάσταση. Δεν έχει νόημα λοιπόν. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την ε, τρομοκρατία όμως, διότι αυτή είναι και μία από τις ε, αιτίες ε, της κατάστασης εκεί. Είναι οι άνθρωποι κατευθύνονται προς την ε, τρομοκρατία και θεωρώ πως τα Ηνωμένα Έθνη είναι υπεύθυνα για την ε, τήρηση της ε, τάξης στην περιοχή. η κυβέρνηση Τραμπ, ο Νετανιάχου, όλοι οι υπόλοιποι φορείς θα συνεχίσουν το παιχνίδι τους εις βάρος των ανθρώπων, όχι μόνο στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά ε, όλη την περιοχή. Όμως πρέπει να βρούμε τρόπους ε, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και ταυτόχρονα Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τα θεσμικά όργανα αλλά και με τα κράτη-μέλη να ασκήσουν πίεση για να αναλυφθούν ανθρωπιστικές ε, ευθύνες στην περιοχή και να μην γίνει έρμεο των ε, συμφερόντων του κάθε ε, κράτους ε, που έχει συμφέροντα στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις για την Γενική ΕΚΟ, άρα λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχετε κάτι να προσθέσετε, κάποια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να το κάνετε. Φυσικά και το θέμα είναι πολιτικό και αυτό βέβαια είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί εντός των πολιτικών ομάδων. Θα ήθελα επομένως να ευχαριστήσω την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να πω ότι η Επιτροπή μας συνεργάζεται με την Ούνρα και με τους άλλους ε, φορείς για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιόρδα της Γάζας. Περνάμε τώρα στο σημείο 20, ανθρωπιστική κατάσταση και εξαναγκαστικός εκτοπισμός στη Βενεζουέλα και άλλες χώρες της περιοχής. Αυτή είναι μια περιοχή του πλανήτη όπου η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται. Το καλοκαίρι άκουσα μάλιστα στο BBC ότι μια γυναίκα μας, που είχε ένα μπαρ στην, ε, στα σύνορα με την Κολομβία έλεγε ότι φτάνουν άνθρωποι στο κατάστημά της ε, πεινασμένοι και πως η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Ε, δεν θα πω όμως περισσότερα διότι υπάρχουν συνάδελφοι εδώ που πήγαν στη Βενεζουέλα και κατ' θα δώσω το λόγο στην Διτζιέκο, αφού ακούσουμε την ε, Τερέζα Χιμένες, ε, διότι πρέπει να φύγει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συναδέλφους που μου έδωσαν το λόγο. Θα ήθελα να μιλήσω ισπανικά και να πω το εξής. Η ανθρωπιστική κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα είναι κάτι το εξωπραγματικό. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είπε ότι είναι η μεγαλύτερη έξοδος που έχει γίνει ποτέ. Μιλούμε για 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, ανθρώπους που φτάνουν στο Περού, στην Κολομβία, στη Βρεζιλία, στον Ισημερινό Υπάρχουν ήδη περιπτώσεις ε, ξενόφοβων περιστατικών στα σύνορα με τη Βραζιλία. Υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή των προσφύγων της Βενεζουέλας. Βλέπουμε απίστευτες περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα είναι σαφές ότι ε, μιλούμε για ανθρωπιστική κρίση η οποία προέρχεται από μια πολιτική κρίση στην οποία δεν βλέπουμε έξοδο γιατί όλες οι, όλα τα ψηφίσματα και οι εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της διεθνούς κοινότητας δεν την χάνουν ε, υποδοχής, δεν τις ακούει κανείς, δεν τα ακούει κανείς. Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας είπε ότι στη Βενεζουέλα δεν υπάρχει πείνα, δηλαδή από τη στιγμή που η κυβέρνηση αρνείται την κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα αυτή, ενώ εμείς βλέπουμε φωτογραφίες ε, γυναικών άνω των 70 ετών να περνούν τα σύνορα κρατώντας το χέρι τους μικρά παιδιά και βλέπουμε ανθρώπους σκελετωμένους από την πείνα, φωτογραφίες ανθρώπων σκελετωμένων από την πείνα ε, που προέρχονται από μια πλούσια χώρα που αντιμετωπίζει μια απίστευτη κατάσταση. Όλα αυτά είναι αδύνατο να κρυφτούν τώρα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα μέσα επικοινωνίας, παρόλο που η κυβέρνηση της Βενεσουέλας προσπαθεί να τα κρύψει. Δεν είναι μόνο ανθρωπιστική η κρίση, είναι ότι δεν μας επιτρέπουν να τους δώσουμε χρήματα, δεν μας επιτρέπουν να μιλήσουμε με την Αντιπρόεδρο. Ε, και θα πρέπει η Κομισιό να μας πει ε, πώς θα φτάσουν αυτά τα χρήματα και πρέπει να τελειώσουμε με τη ρίζα του προβλήματος, να την εξαλείψουμε, γιατί δεν θα συνεχίσουμε να στέλνουμε χρήματα ε, για να κατασπαταλούνται στη συνέχεια με μη επαρκή τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε τα χρήματα για να βοηθήσουμε τα θύματα, αλλά Χρειαζόμαστε πιο ισχυρή θέση να εντείνουμε τις κυρώσεις ενάντια σε αυτό το πολιτικό καθεστώς το οποίο προκάλεσε οικονομική, κοινωνική, ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγούμενο. το οποίο απειλεί όχι μόνο τη Βενεζουέλα, αλλά απειλεί να διαταράξει την ισορροπία ε, τη Νοτιού Αμερικής και αυτής τη πλευρά του πλανήτη μα. Λύστο, συγγνώμη, πρέπει να φύγω και αφήνω ε, το λόγο στους συναδέλφους και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας από εδώ και θέλω να εκφράσω τη θερμή μου στήριξη στην κοινότητα ε, των Βενεζολάνων που ζουν στην Ευρώπη, στην Ισπανία, στη χώρα μου και ε, την στήριξή μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι μετανάστες γιατί, γιατί δεν θέλω να νιώθουν μόνοι τους γιατί αυτό που βιώνουν είναι αφόρητο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει η DG ECO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα πάρουν το λόγο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ε, μίλησα με τον Επίτροπο Στυλιανίδη όταν ξεκίνησε η κρίση με ενημέρωση και με προειδοποίηση για το πόσο σοβαρή θα ήταν η κατάσταση και πόσο είχε σοκαριστεί από τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Η κυρία Ιρέν Χορέης, αν προφέρω σωστά το όνομά σας, έχετε το λόγο. thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ που προφέρατε το όνομά μου σωστά, χωρές λέγομαι. Είμαι επικεφαλής ε, του Τμήματος για τη Λατινική Αμερική στη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ και θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας εσάς την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την στάση σας, διότι η Βενεζουέλα βρίσκεται σε πραγματική ανθρωπιστική κρίση. Και αυτό έχει, δεν έχει ακουστεί αρκετά στην Ευρώπη. Επίσης, ε, να σας πούμε πως ε, καλωσορίζουμε την αποστολή σας στη Βενεζουέλα και στις μεθοριακές περιοχές της χώρας. Θα σας ε, παρουσιάσω τρία θέματα. Πρώτον, την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, την ανθρωπιστική κατάσταση στις γειτονικές της χώρες, οι οποίες ε, έχουν ε, επηρεαστεί εντονότατα από τη μαζική εγκατάλειψη της Βενεζουέλας από τους κατοίκους της και τρίτον το τι κάνουμε εμείς. Κατάσταση λοιπόν στη Βενεζουέλα. Για να προσθέσω ε, σε αυτά που είπε η κυρία Μπασερίλ, η κατάσταση είναι απελπιστική. Η Βενεζουέλα είναι μια χώρα πλούσια σε φυσικούς πόρους, ήταν μια από τις σταθερότερες δημοκρατίες στη Λατινική Αμερική και μια από τις πλουσιότερες χώρες επίσης. βρίσκεται υπό διαρκή οικονομική κακοδιαχείριση τα τελευταία χρόνια και έχουν φτάσει σε ένα σημείο που τα δύο τρίτα των κατοίκων δεν μπορούν να αγοράσουν τρόφιμα. Αυτά τα στοιχεία που σας παρουσιάζω ε, προέρχονται από μία εθνική έρευνα του 2017 για τα νοικοκυριά της χώρας. Έχουμε λοιπόν τα δύο τρίτα των ε, κατοίκων αν μην μπορούν να αγοράσουν τρόφιμα, υπάρχει πρόβλημα υποσυτισμού για το 16% του πληθυσμού είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. 2 εκατομμύρια παιδιά βρίσκονται εκτός σχολείου, δεν έχουν ε, φαγητό, αρκετό ρούχα, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεταφορές. Ε, τα νοσοκομεία κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά διότι δεν έχουν εξοπλισμό, δεν έχουν προϊόντα, φάρμακα και πολύ συχνά δεν έχουν ούτε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Ο πληθωρισμός λοιπόν ε, με δεδομένων όλων αυτών έχει εκτοξευθεί τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Έχει φτάσει σε σημείο που ένας ε, ολόκληρος μισθός ίσα που φτάνει για να αγοράσει κάποιο τρόφιμα για την οικογένειά του για μία εβδομάδα. Υπάρχουν επιχορηγήσεις και κουπόνια για τρόφιμα τα οποία μοιράζονται από την κυβέρνηση και τον τελευταίο μήνα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ιδιαίτερα λόγω της ε, υποτίμησης του νομίσματος της χώρας. Ε, μετά από το πακετάσο, έτσι το ονομάζει, το οικονομικό πακέτο παρουσίασε ο πρόεδρος Μαδούρο και το νόμισμα κατέρευσε λοιπόν, χρησιμοποιεί τα νοικοκυριά και τα, τις τελευταίες τους οικονομίες. Όπως σας είπα, τα δύο τρίτα δεν μπορούν να αγοράσουν τρόφιμα. Φανταστείτε τι θα γίνει στο τέλος της χρονιάς, πόσο θα αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν ε, η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε μαζική εγκατάλειψη της χώρας. αρχικά η έφευγε η μεσαία τάξη, η πιο εύπορη κάτοικοι. Τώρα όμως από τις αρχές του έτους οι φτωχοί και οι ιδιαίτερα φτωχοί είναι αυτοί που φεύγουν από τη χώρα. Και μάλιστα από τα στοιχεία που έχουμε, περίπου 1,5 εκατομμύριο έχει φύγει τον τελευταίο χρόνο. Τα σύνορα με την Κολομβία έχουν υπερχιλήσει. Υπάρχουν χιλιάδες ε, ανθρώπων που φτάνουν κάθε μέρα στα σύνορα με την Κολομβία. Προσπαθούν να βρουν διάφορους τρόπους να επιζήσουν. Ε, πολλοί από αυτούς διασχίζουν τα σύνορα κάθε μέρα για να δουλέψουν και έχουμε 6 εκατομμύρια ε, κάρτες για διασυνοριακές διελεύσεις που έχουν εκδώσει αρχές των δύο χωρών υπάρχουν οικονομικοί πρόσφυγες από την Βενεζουέλα στην Κολομβία. Τετρακόσχες χιλιάδες. Και επιτρέψτε μου τώρα να σας δώσω μερικά στοιχεία για τη μετανάστευση. Επίσημα λοιπόν στην Κολομβία έχουν καταγραφεί 900.000 κάτοικοι ε, της ε, υπήκοη Βενεζουέλας, εκτός από το 1 εκατομμύριο που ήδη είναι στη χώρα. Για το Εκουαδόρ τώρα. Στο Εκουαδόρ το 2018 μόνο ε, έλαβαν χώρα 547.000 ε, είσοδοι στη χώρα. Υπάρχουν περισσότεροι υπήκοοι Βενεζουέλας οι οποίοι είναι επίσημα αναγνωρισμένοι ως πρόσφυγες του Εκουαδόρ. και περισσότερες νέες ε, είσοδοι στη χώρα περνούν, διέρχονται από το Εκουαδόρ για να πάνε στο Περού και τη Χιλή. Ε, το Περού είχε χιλιάδες εισόδους το 2018 και αναμένονται περισσότερες. Μετά, η Χιλή. 150.000 νέες αφήξεις το 2018. 100.000 βρίσκονται ήδη εκεί. Στη Βραζιλία 70.000 αφήξεις φέτος. Στο τέλος του 2017 οι γειτονικές χώρες καλωσόρισαν τους Βενεζουελάνους. και προσαρμόστηκαν, προσάρμοσαν το, την ομοθεσία τους αν θέλετε. έτσι ώστε να μπορούν να χορηγήσουν ειδικέ θεωρήσεις και άδειες εργασίας ε, σε υπηκόους ε, της Βενεζουέλας που έφταναν στις χώρες τους. Όμως, ε, τους τελευταίους μήνες η μαζική έξοδος από τη χώρα και η μαζική είσοδος στις γειτονικές χώρες έχει ε, αλλάξει τα δεδομένα. Υπάρχει ξενοφοβία, αλλαγή της ε, κοινή γνώμης και οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών βρίσκονται υποποίηση για να διεξάγουν αυστηρότερους σε Αυτή τη στιγμή χρειάζεται διαβατήριο για να μπει ένα υπηκό Βενεζουέλα στι ε, γειτονικέ χώρε. Όμω είναι σχεδόν αδύνατο να βρει να εκδώσει διαβατήριο, διότι δεν υπάρχει ούτε χαρτί, ούτε μηχανήματα για αυτό το σκοπό, ούτε καν ηλεκτρικό ρεύμα. Ε, η λίστα αναμονή λοιπόν ε, είναι πολύ μεγάλη και οι φτωχοί δεν έχουν θέση να... δεν μπορούν να βρουν δυνατότητα να βγάλουν διαβατήριο. Έχει γίνει λοιπόν έκκληση από τον ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες την περασμένη εβδομάδα γιατί στα σύνορα της χώρας εγκλωβίστηκε κόσμος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ φτωχοί και ιδιαίτερα ευάλωτοι ως εκ τούτου. Στην Κολομβία η κατάσταση είναι και εκεί απελπιστική, διότι επειδή δεν υπάρχουν χρήματα για να, για να νοικιάσει κάποιο όχημα ή δικό τους όχημα, πολλοί περπατούν για να διασχίσουν τα σύνορα. Αυτό λοιπόν είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τα παιδιά και τις ε, γυναίκες οι οποίοι είναι εύκολο να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης ε, οικονομικής, σεξουαλικής και γενικότερης εκμετάλλευσης. κατάσταση στις γειτονικές χώρες έχει αποσταθεροποιηθεί, ιδιαίτερα στην Κολομβία και αυτό βάζει σε κίνδυνο την ειρηνευτική διαδικασία που είναι κάτι πολύ εύθραυστο όπως γνωρίζετε. Ορισμένοι νέοι Βενεζουελάνοι στρατολογούνται σε εγκληματικές συμμορίες, σε διακι... Ε, για διακίνηση ναρκωτικών και σε ένοπλες ομάδες στην Κολομβία. Έχει γίνει ήδη αρκετές φορές έκκληση από τις γειτονικές χώρες για την παροχή διεθνούς προς, ε, βοήθειας. Το Εκουαδόρ επίσης έχει ζητήσει Διεθνή Σύνοδο για την ε, αντιμετώπιση της κρίσης στην περιοχή. Τώρα, τι κάνουμε εμείς. Η ομάδα μας ξεκίνησε δράση στη Βενεζουέλα πριν από δύο χρόνια. Αρχικά σε μικρή κλίμακα. Ξεκινήσαμε ε, στηρίζοντας την καριτά της Βενεζουέλας με δράσεις για επιστηστική βοήθεια. Πέρυσι ξεκινήσαμε ε, να στηρίζουμε τον Ερυθρό Σταυρό και σε συνεργασία με την Επατερμοστία για τους πρόσφυγες, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και αρκετές μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αρχίσαμε να δημιουργούμε ένα ανθρωπιστικό δίκτυο στη Βενεζουέλα. Διότι ένα από τα προβλήματα που μας εμποδίζουν στην παροχή βοήθειας είναι ακριβώς ότι επειδή η Βενεζουέλα ήταν πολύ πλούσια χώρα, δεν υπήρχε παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, δεν υπήρχαν ανθρωπιστικές οργανώσεις στη χώρα. Ε, εμείς λοιπόν ε, παρέχουμε βοήθεια, προστασία σε διάφορους τομείς. Μετά την επίσκεψη του Επιτρόπου Στυλιανίδη στη Κολομβία και στα σύνορα έχουμε δεσμεύσει περισσότερα κονδύλια και έχουμε επεκτείνει την προστασία μας εντός της ε, χώρας αλλά και στις γειτονικέ χώρες. Παρέχουμε βοήθεια στην Κολομβία, ιδιαίτερα στις ε, μεθοριακές περιοχές και στις κοινότητες εκείνες οι οποίες φιλοξενούν μεγάλο και αυξανόμενο αριθμό ε, Βενεζουελάνων. Επίσης παρέχουμε βοήθεια στον Ερυθρό Σταυρό στο Εκουαδόρ, όπου έχουν εισρεύσει πολλοί άνθρωποι και χρειάζεται βοήθεια η περιοχή αυτή. Αλλά και στα σύνορα με την Βραζιλία, σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, ε, παρέχουμε βοήθεια. Είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε καταφέρει να παρέχουμε βοήθεια στο εσωτερικό της χώρας, Και γνωρίζουμε φυσικά ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, ποτέ δεν ζήτησε διεθνή ε, βοήθεια. Και οι σχέσεις μας με την κυβέρνηση είναι ε, πολύ λεπτές. Όμως προσπαθούμε να ενεργούμε με απόλυτη διαφάνεια και οι εταίροι μας κατάφεραν να έχουν πάντα την άδεια της, ε, των τοπικών κυβερνήσεων και τη συνεργασία τους ή ε, την ανοχή τους. Ως αντάλλαγμα, εμείς φροντίζουμε πάντα να διατηρούμε χαμηλό χαμηλούς τόνους και να μην εμποδίζουμε το έργο των τοπικών κυβερνήσεων. Φέτος, το Μάιο, συζητήσαμε εντός Γενικής Διεύθυνσης και ε, με άλλους φορείς τη δημιουργία ενός συμφώνου για τη Βενεζουέλα. Η Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΚΟ αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ε, Βενεζουέλα, διότι ακριβώς πρέπει να συνεργαστεί με την ε, κυβέρνηση εκεί. Στην Κολομβία όμως, για να αποκτήσουμε έτσι ένα καλύτερο πλαίσιο, έχουμε καταβάλει προσπάθειες συνεργασίας και δημιουργίας αυτού του δικτύου. Βέβαια, επειδή στη Βενεζουέλα και τις γειτονικές χώρες υπάρχει τεράστια ανάγκη βοήθειας, ε, δεν αρκούν όλα αυτά και πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Εμεί ευχαριστούμε για αυτή την πλήρη ενημέρωση όσον αφορά την εικόνα της κατάστασης. Ναι, τώρα το συζητήσαμε το θέμα και ευτυχώ και από την Επιτροπή. Ε, Ακριβώ είναι φρικτά όλα αυτά τα οποία είδατε. Ε, και οι συνάδελφοι για να μας τα πούν τώρα, αυτοί που τα είδαν, ο κύριος ε, Φαρία και η κυρία Μπεθέρα μετά. Ευχαριστώ πρόεδρε ο Φαρία. Είναι σημαντικό το θέμα. Και να σας πω ότι ήμουν ένα από τα μέλη της αντιπροσωπείας που μετέβη στη χώρα. Πήγα στην Κουκούτα, στα σύνορα με την Κολομβία. Και μπορώ να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο ε, ένας άνθρωπος να δει αυτά τα οποία είδα. Είδαμε ανθρώπους που σκότσαν σε απελπιστική κατάσταση. Αγανακτισμένοι, θυμωμένοι, όπως ανέφερε η Τερέσα. Παιδιά χωρίς τους γονείς τους. Τη νύχτα που πήγαμε εκεί, μας είχαν πει ότι πέθαναν 7 Βενεζολάνοι καθοδόν προς την Κουκούτα λόγω του κρύου. Προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τη χώρα. Ήταν 10 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα και σταμάτησαν να δημιουργηθούν και πέθαναν εκεί. Αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο. Αυτά από πλευράς του τι είδαμε στα σύνορα, γιατί μέσα στη χώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται παρόλα αυτά. Ακούσαμε τι είπε Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ισχύουν φυσικά για το τι γίνεται μέσα στη χώρα. Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όσο ακούσαμε. Πήγα για τις εκλογές στη χώρα το 2015 και από τότε με έχουν ενημερώσει οι Βενεζολάνοι και μου ζητούν να τους βοηθήσουμε. Φάρμακα ζητούν, τρόφιμα, τα πάντα. Αλλά είναι τόσο δύσκολο να περάσει αυτά λόγω του καθεστώτος Μαδούρο. Δεν θέλουν να αποδεχθούν ότι υπάρχει κρίση ανθρωπιστική και αφήνει τον κόσμο στις τύχες του να πεθάνει. Να μην με αλλά μια που πήγα εκεί πρέπει να δώσω τις αρχές Κολομβίας συγχαρητήρια γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο τόσα κάνουν. Είναι καταπληκτικό το έργο του στα σύνορα, αλλά θα πρέπει κάποιες άλλες χώρες Όπω το Περού και ο σημερινό θα πρέπει να ε, επικριθούν γιατί ζητούν από τους πρόσφυγες διαβατήρια. Απαράδεκτο. Πού να βρουν διαβατήριο οι άνθρωποι στη Βενεζουέλα. Αυτό σημαίνει ότι δεν τους αφήνουν να περάσουν. Επίσης να σας πω ότι ανησυχώ και για τόσο γίνεται στη Βραζιλία. Ο κόσμος που φεύγει λόγω των φρικαλαιοτήτων που αντιμετωπίζουν από πλευράς Μαδούρο περνάνε τώρα. Πώς έγινε στη Βραζιλία ευτυχώς Κάποιοι τους υπερασπίζονται στον αγώνα τους να έχουν το δικαίωμα να μπορούν να μείνουν στη χώρα τους, αλλά Τέλος πάντων, μπράβο για την πρωτοβουλία, Πρόεδρε. Θα ε, πρέπει να πιέσουμε την κυρία Μογγυρίνη. Όπως είπε η Τέρεσα, να πιεστεί περισσότερο η κυβέρνηση. Να πιέσουμε για κυρώσεις. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι Βενεζολάνοι είναι πρόσφυγες. Αυτό θα κάνει μεγάλη διαφορά. Ο κόσμος κάθε μέρα πεθαίνει. Στη χώρα. Και σας ευχαριστώ. Αυτό κάπως μου θυμίζει, λέει ο Πρόεδρος. Στο παρελθόν ότι έχει αυτό ξαναγίνει. Θυμάμαι το Σεπτέμβριο στην Τουρκία, πριν τη μαζική έξοδο του κόσμου της περιοχής προς την Ευρώπη. Και όπως είπατε, κάποιοι είχαν μαζί τους κάποια χρήματα, βοηθήσαν την οικονομία και ήταν και κάποιοι άλλοι μετά που θέλαν βοήθεια, ένα σωρό προβλήματα. Ήταν πιο φτωχοί, πιο δύσκολο. Άρα πρέπει να προγραμματιστούμε. Τι θα κάνουμε, ίσως για αυτό την κατάσταση να κάνουμε κάτι στην Ολομέλεια. Να το συζητήσουν τα, οι πολιτικές ομάδες την επόμενη εβδομάδα. Η κυρία Μπεθέρα που ήταν στην αντιπροσωπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή για το έργο της και για την ενημέρωση. Να το τι μπορούμε να κάνουμε. Να θυμηθούμε τι έλεγε στο εξώφυλλο και τι έλεγε μέσα. Το time από καμιά διετία ήταν μια σπόμενη φωτογραφία τρομερή και έλεγε ότι πρόκειται για ολοκληρωτική κατάρρευση της χώρας. Ότι πεθαίνει η χώρα. Πέρασαν δύο χρόνια. Δεν πρόκειται απλώς για κατάρρευση. Τα πράγματα χειροτέρευσαν πρόκειται για κάποια ρητή, ξεκάθαρη πολιτική απόφαση δεν χωρούν δικαιολογίε. Ούτε πρόκειται για θεομηνία, ούτε για πόλεμο. Που να εξηγεί γιατί αυτά τα 30 εκατομμύρια του κόσμου σε μια πλούσια χώρα εδώ και τόσα χρόνια ζουν μέσα στην φτώχεια, την ανέχεια, την πείνα. Δεν έχουν τα βασικά μέσα. Και αυτά, αυτή, η έλλειψη χρησιμοποιείται από το καθεστώς του Μαδούρου ως όπλο. Είπαμε για τις ατομικές κυρώσεις της Ευρώπης, αλλά, αλλά συστηματικά για την καταστολή, για την καταπίεση του κόσμου, για τη διατήρηση στην κυβέρνηση, στο διαφθαρμένο καθεστώς τα χρησιμοποιούν όλα αυτά. Και είχαμε ανακοίνωση του, του ΙΕ που έλεγε για τα 2 εκατομμύρια που φεύγαν, τώρα είναι 4 εκατομμύρια. Κάθε, κάθε μέρα περνάνε την γέφυρα στα σύνορα χιλιάδες. Αυτοί που μπορούσαν. 10-15% του πληθυσμού σχεδόν. Τώρα αποτελούν την διασπορά του λαού σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι θεομηνία ούτε πόλεμο, επαναλαμβάνω. Εμείς που πήγαμε εκεί τέλη Ιουνίου εκεί στην Κουκουτά, στην γέφυρα Μπολίβαρ, είδαμε λάβοντας υπόψη ό,τι έχουμε δει κινήσεις, φτωχούς ε, προσφυγιά όλο αυτό που είδαμε εκεί δεν έχει καμία σχέση με ό,τι είχαμε δει προηγουμένως πρόκειται για ένα ανθρώπινο ποτάμι τρομερών διαστάσεων αυτό έγινε στο Σουδάν, μπορεί κανείς να καταλάβει τι γίνεται, αλλά στη γέφυρα κούκουτα και στα άλλα συνοριακή της χώρας δεν καταλαβαίνεις. Είναι πολύ χειρότερα. Επομένως τώρα, επί του πρακτέο τι μπορούμε να κάνουμε ως Ένωση. Ακριβώς όπως τα είπατε, μέσα στη χώρα μπορούμε μόνο κρυφά να παρέμβουμε γιατί το καθεστώς θέλει να αποκλείσει κάθε δυνατότητα επιβίωση για τον κόσμο, αλλά δεν μπορεί να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια. Όπως είναι επομένως τα πράγματα, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα στα σύνορα. Ε, είναι σημαντικό να το κάνουμε με διαφάνεια, ε, με προσοχή, ούτως ώστε να πιάσουν τόπο τα λεφτά. Το, το φαγητό είναι πολύ σημαντικό, η θυσιμότητα η παιδική είναι φρικτή. Όλες, όλες οι κοπέλες που να γεννήσουν φεύγουν από τη χώρα. Καμία δεν γεννάει στη Βενεζουέλα. Πολλές φορές φυσικά είναι αθέλητη η κοίηση. Επομένως είναι πρόβλημα μεγάλο το θέμα της διατροφής, της υγιεινής υπάρχουν ε, πάρα πολλές ασθένειες που ξεσπούν και όπως είπαμε βοηθάει η Κολομβία όλες τους φεύγουν μπράβο για τη διαχείρισή τους δείχνουν επαγγελματικότητα συνέπεια για αυτό το φαινόμενο και όλοι οι Κολομβιανοί με τους οποίους μίλησαμε μας μίλησαν για τους αδερφούς Βενεζολάνους γι' αυτό σας λέω υπάρχουν ανάγκες σε τρόφιμα για βασική υγιεινή μέρες περπατάνε οι οικογένειες για να φύγουν δεν έχουν ηλεκτρισμό Είχαμε μια ολόκληρη περιφέρεια που δεν είχε ηλεκτρισμό, δεν είχε ρεύμα. Πλημμύρε. Μιλάμε για χρόνια που έχουν πληγεί πολλές περιφέρειες από πλημμύρες. Γι' αυτό σας λέω. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και αποτελεσματική την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά από την άλλη μεριά να είμαστε αυστηροί, κατηγορηματικοί από πλευρά πολιτική τοποθέτηση. Είπαμε πώς αντιδρούν τα κράτη της περιοχής, από πλευρά σταθεροποίηση και σταθερότητα της περιοχής. Άρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κάποια εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι το σωστό, κατά τη γνώμη μου και έτσι να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι ναι, κάτι μπορεί να γίνει. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Θέλει άλλο το λόγο. Ο Σάρλ. Ναι. Όσοι ήταν τόπου, τι πιστεύουν. Μπορεί κάτι να δράσει μέσα από τις τοπικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται είναι αυτό εφικτό. Τον Ερυθρό Σταυρό, την Κάριτας, άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Η κυρία Μπεσέρα μας είπε ότι είναι δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να δράσει κανείς από έξω. Άρα υπάρχουν διάμεση φορείς που δραστηριοποιούνται επί τόπου και που μας επιτρέπουν να τους διοχετεύσουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Mm Με άλλα καθεστώτα, στη Βόρεια Κορέα για παράδειγμα, υπάρχουν τοπικές οργανώσεις εκεί και μπορεί κανείς να τις εμπιστευθεί. Αυτό ρωτάω. Τώρα, ένα συμπληρωματικό ερώτημα. Η τοπική φορείς είναι αρκετά αξιόπιστη? Η βοήθεια που θα διοχετεύουμε στη Βενεζουέλα θα φτάσει στα σωστά χέρια. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει η Πρόεδρος, ότι συνεργάζεται με την Κάριτας, αλλά ε, θα σας ξανδώσουμε το λόγο να μας τα εξηγήσετε. Συγκεντρώνουμε τώρα τις ερωτήσεις, τις σημειώνετε και απαντάτε ομαδικά στο τέλος. Ο Ευχαριστώ, ευχαριστώ για το ερώτημα αυτό. Ναι, υπάρχουν τοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται επί τόπου. Αλλά δεν πρέπει να τους πούμε ποιοι είναι, γιατί θα έχουν πολλά προβλήματα με το καθεστώς Μαδούρο. Το που μας είπαν είναι ότι υπάρχουν άτυποι διάδρομοι ανθρωπιστικής στήριξης, αλλά δεν είναι αυτό επίσημο και πρέπει έτσι να μείνει, με άτυπο τρόπο. Δεν μπορώ να σας πω ποιος μας το είπε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν μέσα, αλλά πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Είναι ένα σύστημα εξαιρετικά περίπλοκο γιατί και οι αρχές οι επίσημες της Βενεζουέλας γνωρίζουν ότι υπάρχουν άτυποι διάδρομοι παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και χρεώνουν. Πρέπει να παραμείνει δηλαδή άτυπη και ανεπίσημη η οδός. Αλλά υπάρχουν φορείς με τους οποίους μπορούμε να είμαστε σε επικοινωνία. και προσπαθούμε να τους δώσουμε με άτυπο τρόπο τα αγαθά που χρειάζονται. Όχι είναι η απάντηση στο ερώτημα εκτός μικροφώνου του Σάγλα. Η πρόεδρος. Είχαμε ψήφισμα τον Ιούλιο για τη Βενεζουέλα, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Είχαμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό. Δεν υπάρχουν νεότερα για το θέμα των διαβατηρίων. Για το θέμα των διαβατηρίων στις γειτονικές χώρες θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή στο τέλος. να δούμε πώς μπορούμε να μιλήσουμε με τις άλλες χώρες για το θέμα των διαβατηρίων. Για την έκδοση των διαβατηρίων θα μας ζητήσουν να δώσουμε περισσότερη βοήθεια ε, ως αντάλλαγμα για την έκδοση αυτή. Ο κύριος Κορνιά όμως θα ήθελα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι διπλωματική φύσεως η ερώτησή μου. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ασκεί περισσότερη πίεση στην Βενεζουέλα και γιατί δεν αναζητά τον συντονισμό, δεν επιδιώκει τον συντονισμό των ευρωπαϊκών χωρών. Όλοι ξέρουν ότι το καθεστώς Μαδούρο είναι διεφθαρμένο καθεστώς. Και το χαρακτηριστικό των διεφθαρμένων είναι ότι δεν κρατούν τα χρήματά τους στην πατρίδα τους. Άρα έχουμε και έναν άλλο τρόπο, μία άλλη διαβλό για να ξεκινήσουμε σοβαρές συζητήσεις με την ε, κυβέρνηση. Είναι πράγματι πάντοτε βρίσκονται ε, χρήματα σε κάποια τράπεζα σε κάποιο μέρος του κόσμου, η Να προσθέσω κάτι που διαφωτίζει τη συζήτηση, πιστεύω. Η Οργάνωση Αμερικανικών Κρατών πρότεινε και έγινε έκθεση από τρεις εμπειρογνώμονες για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί στη Βενεζουέλα και έχουν ταυτοποιηθεί και αναγνωριστεί 7 εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από το καθεστώς Μαδούρο και το πιο σοβαρό από όλα είναι αυτό που έχει να κάνει με τη χρήση της πείνας και της φτώχειας ως εργαλείο καταπίεσης και καταστολής. Αυτή η έκθεση παρουσιάστηκε εδώ από τον Άριφιν Κότλερ, πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης του Καναδά και είναι αρκετή βάση ώστε οι χώρες που έχουν υπογράψει τη χάρτα της Ρώμης να προσφύγουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να ξεκινήσει τη διερεύνηση για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Βενεζουέλα τα οποία δεν παραγράφονται. Και αυτό είναι κάτι που μπορούν να κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή κατά την οποία έχουν επιβεβαιώσει την απόφασή τους να προχωρήσουν και να ανοίξει φάκελος ε, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Το έχουν κάνει τέσσερις χώρες, το, Περού, η Κολομβία, η Χιλή και ίσως και η Παραγουάη. Ο Καναδάς στηρίζει σαφέστατα, δεν το έχει βέβαια πει ξεκάθαρα, αυτή τη διαδικασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης και θα πρέπει να ενισχύσουν οι ευρωπαϊκές χώρες τη θέση αυτή γιατί είναι μια θέση απολύτως αντικειμενική. Η έκθεση βασίζεται σε εκατοντάδες καταγραφές ανθρώπων βασανισμένων. Δεν μιλώ μόνο για πείνα και λοιμό, αλλά και για βασανιστήρια σωματικά, σεξουαλικά, τα οποία συστηματικά έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένας πολύ συγκεκριμένο τρόπος δράσης αυτός θα πρέπει να δουλέψουμε για να ξαναμπεί η Βενεζουέλα στο σωστό θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει να δουλέψουμε για να ανοίξουμε ένα διάβλο παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, θα πρέπει όμως και να δράσουμε ενάντια των υπευθύνων και το, ο τρόπο αυτό ταιριάζει στην αρμοδιότητά μας. Δηλαδή να ζητήσουμε από το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο τη Χάγης να διερευνήσει τα αδικήματα, παράλληλα με τι λοιπέ μα δράσει. Ω, σε παρακαλώ. Νομίζω ότι σήμερα θα είμαι πολύ σύντομος. Νομίζω ότι προς το παρόν πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ούτε το Βατικανό δεν μπορεί κάτι να κάνει. Είναι όλα μπλοκαρισμένα. Και κρίμα που το λέω, αλλά η μόνη λύση είναι να περάσουμε από την Κούβα. να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις διπλωματικές με τους Κουβανούς για να φέρουν αυτοί κάτι στη Βενεζουέλα. Να δώσουν αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια. Μόνο έτσι γίνεται. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και εντάξει, πρέπει όντως να σταθούμε και στη Χάγη να πάμε αλλά να στείλουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Γιατί οι πολίτες μας ρωτούν κάθε μέρα, μα τι κάνετε εκεί, εκεί πεθαίνει ο κόσμος. Εσείς κάνετε διακοπές, έχετε διακοπή της, των κοινοβουλευτικών εργασιών τον Αύγουστο και τι κάνετε και εκεί πεθαίνει ο κόσμος. Γι' αυτό κυρία Πρόεδρε σας χαίρομαι που κάνετε αυτή τη συζήτηση σε μια τόσο επίκαιρη χρονική στιγμή. Σας ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην DG ECO. Uh, να σας δώσουμε τώρα το λόγο, να μας πείτε ό,τι άλλο χρειάζεται. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω για την περιοχή της κατάστασης, όπως τα ακούσαμε. Απελπιστική η κατάσταση. Το Κοινοβούλιο το πήγε πάρα πολύ καλά με την αποστολή. Ζητήσατε να σα ενημερώσω για το τι καινούργια στοιχεία υπάρχουν. Υπάρχουν τα εξή δύο. Πρώτα-πρώτα έχει αυξηθεί ο πληθωρισμό και πρόσφατα είχαμε ένα πακέτο οικονομική μεταρρύθμιση που αποστέρισε τελείω από αγοραστική δύναμη τον κόσμο. Επομένω έχουμε μεγάλη υποτίμηση και επίση μεγάλη αύξηση στι ε, τιμέ βασικών ειδών επίσης μείωση επιδομάτων και όσοι είχαν κάποιες αποταμιεύσεις τις χάσανε. Οπότε μιλούμε για τα δύο τρίτα του κόσμου που δεν μπορούν να αγοράσουν το καθημερινό φαγητό, στο πράγμα ακόμα γεροδοσμωματικότητα και γι' αυτό αυτό προκάλεσε καινούργιο ρεύμα εξόδου. Και αν τα στοιχεία είναι αυτά τα οποία τώρα ακούσαμε και ήταν απελπιστικά, ε, εγώ νομίζω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι πάνε στις ε, ιδανικές χώρες είναι ακόμα περισσότεροι. Οπότε γι' αυτό το λόγο και σφίξαν τους ελέγχους τους συνοριακούς οι κοινωνιάζουσες χώρες. Α, για το Περού ξέρω δύο πράγματα. Υπάρχει εκεί κάποιο είδους βίζα ανθρωπιστική που την θεσπίσανε ειδικά για τους Βενεζολάνους και τους επιτρέπουν να έχουν πρόσβαση στο να βρουν δουλειά, σε κάποιες βασικές υπηρεσίες. Πάντως έκαναν αυστηρότερες προϋποθέσεις για είσοδο στη χώρα. Τους ζητάνε δηλαδή διαβατήριο και κάποιο ποσό σε δολάρια. Δεν τα έχει αυτά ο κόσμος και για να βρουν τα χρήματα εκπορνεύονται, μου τα λένε αυτό με το, για το Εκουαδόρ γίνεται αυτό. Μπαίνουν σε λεωφόρια να πουλήσουν ό,τι ό,τι υπάρχοντα έχουν. Δηλαδή πολύ περισσότεροι αυτοί που θέλουν να ξεπουλήσουν ότι έχουν παρά οι επιβάτες και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένταση, υπάρχουν συγκρούσεις ε, και εχθρικό κατά αυτών των ανθρώπων. Έρχονται με τα, πόδια, εκπορνεύονται, αποτελούν για τους άλλους γείτονες φτωχούς ε, ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας. Κάνουν ό,τι μπορούν για να επιβιώσουν στα όρια της νομιμότητας. Ε, υπάρχει θέμα ασφάλειας και έτσι και η Βενεζουέλα πάντοτε δεν είχε μεγάλη ασφάλεια, πάντοτε είχε μεγάλη εγκληματικότητα. Οπότε τώρα αυξήθηκε η εγκληματικότητα λόγω των ελλείψεων σε κάθε είδος. Όλο ένα και λιγότερη ασφάλεια στη χώρα. Να πως έχει το τοπίο. Σας ευχαριστώ γιατί είναι σημαντικό το να δείχνετε ενδιαφέρον γιατί έτσι μας βοηθάτε να προσπαθήσουμε καλύτερα, να προσπαθήσουμε περισσότερο και τελικά να κινητοποιήσουμε περισσότερους πόρους. Τώρα, για αυτά που ρωτήσατε, με ποιον συνεργαζόμαστε. Υπάρχει δίκτυο ΜΚΟ. Ε, στη χώρα πάντοτε ήταν μικρής κλίμακας. Προσπαθούμε εμείς να ενισχύσουμε το κύκλωμα αυτό και τώρα συνεργαζόμαστε με την τοπική κάριτας, Ερθρό Σταυρό, την οργάνωση ΦΕ Αλεγρία, που υπάρχει σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής και καταφέραμε έτσι να έχουμε μία μόνιμη παρουσία στη χώρα. Οπότε έχουμε κάποιους ε, ειδικού που παντρώνουν ένα γραφείο στην Πογκότα και πηγαίνουν έρχονται επίσης. Κάποιους ειδικού που εκεί είναι μόνιμα εγκατεστημένοι και επιβλέπουν τη ΜΚΟ για τον ΟΗΕ, υπάρχει ο IOM, η UNICEF, ο UNHR και όλοι αυτοί είναι εκεί και επίσημα παρά όλες τις δυσκολίες ε, παράγουν έργο στη χώρα. Θέλουμε επομένω να στηρίξουμε τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού δικτύου. Να υπάρξει συντονισμός των προσπαθειών. Ναι, ναι, αλήθεια είναι όλα που ακούσαμε για τις δυσκολίες. Αλλά δεν θα πρέπει να κάνουμε πίσω. με τον οργανισμό πάχο φροντίζουμε να υπάρχουν φάρμακα ό,τι ό,τι μπορούμε να καταφέρουμε. Πολλές φορές σε επίπεδο τοπικών αρχών τα πράγματα είναι ευκολότερα γιατί και οι τοπικές αρχές είναι σε απελπιστική κατάσταση. Η αξιοπιστία, όπως το λένε στα αγγλικά, των ε, οργανώσεων, οργανισμών αυτών. Δεν είναι τόσο ισχυρή αυτή η φορής και ένα από τα προβλήματα είναι ότι το προσωπικό συνέχεια αναλάσσεται γιατί ο κόσμος φεύγει. Η κάρτα ας πούμε, είχε κάποιους γιατρούς, οι γιατροί φύγανε από τη χώρα. Τα συνέχεια θα πρέπει κανείς να εκπαιδεύει, να ξαναεκπαιδεύει για να επανδρώσει τον οργανισμό ε, και να υποπτεύσει. Νομίζω ότι τα καταφέρουμε πάντως. Παρά όλα αυτά τα σημεία που είπατε ότι πρέπει να προσέξουμε έστω και ανεπίσημα. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που ήθελα να σας πω. Για τον ΟΗΕ επίσης και στο μέτωπο της μετανάστευσης και η UNHCR και ο Οργανισμός Μετανάστευσης ε, ασχολούνται εντατικά σε όλες τις ε, γειτονικές χώρες. Ε, έχουν απευθύνει κάποιες εκκλήσεις κατεπίγοντα χαρακτήρα ο IOM και η UNHCR 32 εκατομμύρια έχουν διατεθεί Δεν έχουμε και μεγάλη πρικοδότηση για την περιοχή πάντως, γιατί όπω είπαμε στην αρχή θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα. Υπάρχει η ομάδα εργασία Κόλακ του Συμβουλίου. Κάθε μέρα, μάλλον κάθε εβδομάδα τέλος πάντων συζητούν για την Βενεζουέλα. σίγουρα και στην εξωτερική υπηρεσία ασχολούνται, θα μπορούσαν να έρθουν συνάδελφοι να σας τα πούν εδώ, δεν μπορώ να σας τα πω εγώ. Πάντως η Ένωση έχει προσπαθήσει για διαμεσολάβηση, έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες συνεννόησης ε, ε με την αντιπολίτευση, το θέμα επίσης των ατομικών ε, ε, κυρώσεων ε, σε σχέση με πολιτική βία. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες γιατί εγώ ασχολούμαι με τα ανθρωπιστικά στην ΕΚΟ. Όπως προείπα, οι γειτονικές χώρες πιέζονται και από πέρσι συγκρότησαν την ομάδα Λίμα. Αυτή η ομάδα υπάγεται στον φορέα των λατινοαμερικανικών χωρών. Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στη Βενεζουέλα Και ο Καναδάς συμμετέχει σε αυτή την ομάδα, αλλά όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι παρατηρητής. Έχουν απευθύνει διάφορε εκκλήσει αύξηση τη ανθρωπική βοήθεια ή τη ομάδα αυτή. Οπότε στο μέλλον τι θα κάνουμε. Θα βοηθήσουμε σε σχέση με το μεταναστευτικό εκεί όλους αυτούς τους ευάλωτους, αυτούς όλους που είναι παγιδευμένοι ούτως υπήνουν στα διάφορα σύνορα. Όλους αυτούς που είναι στόχος ε, εκμετάλλευσης. Και επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσέξουμε να παράσχουμε ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στη χώρα. Να αυξήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στη χώρα. Να σταματήσει να πεθαίνει ο κόσμος και να φεύγει μαζικά. Γιατί αυτή η έξοδος είναι κακή και για αυτούς που παραμένουν στη χώρα. Αν φύγει ο θείος, ο ο γιος που είναι ακόμα σε ενεργή ηλικία, αυτοί οι οποίοι μένουν πίσω είναι οι ανήλικοι, γιαγιάδες, οπότε και αυτοί βρίσκονται σε δύσκολη θέση έτσι. Και πάλι σας ευχαριστώ που μας καλέσατε και ό,τι χρειάζεστε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκαμε το χρόνο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι ένα θέμα που το συζητήσαμε τον ε, μήνα που μας πέρασε, οπότε νομίζω πως είναι λίγο νωρίς να ζητήσουμε να συζητηθεί πάλι στην Ολομέλεια. Μπορούμε να στείλουμε μια επιστολή στην ε, κυρία Μογκερίνη, να πούμε ότι θέλουμε να συζητηθεί, ότι ε, είμαστε αποφασισμένοι να ασχοληθούμε με το θέμα ενεργά και μετά να τη ζητήσουμε να εντείνει το διάλογο με τις γειτονικέ χώρες για να ανοίξουν το, να, να κάνουν πιο εύκολη την έκδοση θεωρήσεων για να βρεθεί κάποια λύση διότι είναι πολύ δύσκολο να μπει βοήθεια μέσα στη Βενεσουέλα, έτσι θα πρέπει τουλάχιστον ο κόσμος να μπορεί να βγει, να, να τραφεί, να μην πεθάνει από την πείνα. Ε, είναι τραγικό, είναι κάτι που μας σοκάρει ότι η Βενεζουέλα, μια τόσο πλούσια χώρα, ε, περνά τέτοια κρίση. Που όμοιά τη ε, δεν υπάρχει ούτε σε μερικές από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Μας λένε ότι είναι από τις χειρότερες περιπτώσεις που έχουν δει, διότι οι υποδομές ε, έχουν πρόβλημα. Θα... Ήταν καλό λοιπόν να ζητήσουμε από τον ε, Γενικό Γραμματέα να στείλει μια επιστολή και μετά να αναλάβουν οι συντονιστές. Ίσως ε, καλό θα είναι να περιμένουμε, να αφήσουμε ανοιχτό διεύλο επικοινωνία με τη Γενική Διεθνή ΕΚΟΤΣΙ, ώστε αν δεν γίνει τίποτα να επαναλάβουμε τις εκκλήσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και ε, συνεισφέρατε με την εμπειρία σας. Ε, το σημείο 21 είναι η ώρα των ερωτήσεων. Δεν υπάρχει κάποια σχετική ερώτηση. Το 22 διάφορα. Δεν έχω σημειώσει ότι υπάρχει κάποιο θέμα στα διάφορα. Επόμενη συνεδρίαση. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Τζόζεφ, πριν φύγεις. την επόμενη φορά που θα καλέσουμε πρέσβεις από άλλες χώρες, ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να έρθει και ε, ο πρεσβής της Βενεζουέλας έτσι σε μια μικρή συνεδρίαση για να μας ενημερώσει. Ε, προσεχή συνεδρίαση 24 Σεπτεμβρίου 2018 από το, τις 2.30 και αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τους διερμηνείς.